Okay, colleagues, if I can reconvene the meeting and I'll start by... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε τη συνεδρίασή μας και την αρχίζουμε με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών που κάναμε σήμερα το πρωί. Οι συγητές καταρχάς, τρεις κυρίες εκθέσεις από την Επιτροπή των Μεταφορών. Κανονισμός για τους περιοδικούς ελέγχους των ε, οχημάτων με κινητήρα. Μετά έχουμε τον έλεγχο των εμπορικών οχημάτων και πρόταση οδηγίας τρίτων για τροποποίηση της 3799 για την καταχώρηση, έγραφα καταχωρήσεως ε, οχημάτων. Και αποφασίζουν οι συντονιστές τρεις εκθέσεις να γίνουν με ένα στην όμως σχετική απόφαση αποφασαδής για το σε ποιον θα ανατεθούν να, να αναβληθεί την προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών 17 Σεπτεμβρίου. Και εκεί θα αποφασιστεί ποιο θα βλέπει. Μετά έχουμε έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση της οδηγίας για την ε, περιοδική κατάρτιση των οδικών οχημάτων μεταφορά επιβατών και είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλία. Περιμένουμε όμως το 17 Σεπτεμβρίου και πάλι για να δούμε κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς μιας ομάδας για την ανάθεση της έκθεσης. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα το αφήσουμε. Στη συνέχεια έχουμε την ε, έκθεση για την υλοποίηση του κανονισμού 2008 για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία με απόφαση να μην αναλάβουμε δράση και στην ανάπτυξη της αγοράς των σιδηροδρόμων αποφασίστηκε να μην αναλυφθεί δραστηριότητα προς το παρόν αλλά να αξιοποιηθεί η εν λόγω έκθεση ως έγγραφο αναφορά για την αναθεώρηση, την εξέταση μάλλον του τετάρτου πακέτου για τους συντροδρόμους. Γνωμοδοτήσεις τώρα είχαμε πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού 443-2009 για τον προσδιορισμό των ε, διατυπώσεων για την επίτευξη των προποθέσεων για την επίτευξη του στόχου μείωση του εξτίου του άνθρακα για τα νέα επιβατικά θετικά αυτοκίνητα το 2020 με αρμόδια κατ' ουσίαν την Επιτροπή Περιβάλλοντος και απόφαση ένας εισηγητής να αναλάβει για το θέμα αυτό και για το θέμα της εναλλαγής, rotation δηλαδή, και αυτό η ομάδα να είναι από, ο εισηγητής να είναι από τους, από τους σοσιαλιστές δημοκράτες. Είπαμε επίσης ότι στις 13 ε, Σεπτεμβρίου περιμένουμε προτάσεις ε, για το 2013-2013. Είχαμε δύο προτάσεις για επισκέψεις ε, στην ε, βόρεια, Δυτική Αγγλία και άλλη μία για τη Washington της ΗΠΑ. Άλλες δύο προτάσεις για επισκέψεις κατατέθηκαν επίθεση. Πάντως λέμε ότι οποιασδήποτε άλλες προτάσεις και για επισκέψεις και για ακροάσεις, για σχόλια θα πρέπει να αφορούν τις ημέρες των Επιτροπών. Αυτά μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων για επίσκεψη αντιπροσωπιών μας στο εξωτερικό. Όπως είπα, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου προτάσεις για επισκέψη στο εξωτερικό ή ενδεχομένως ακροάσεις σε θέματα διατλαντικής συνεργασίας. Αποφασίζουν οι συντονιστές να, προσκαλέσουν, να καλέσουν τους συναδέλφους της Επιτροπής των Μεταφορών για κατάθεση προτάσεων τροπολογιών απευθείας στην έκθεσή της για τις διατλαντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι. Επίσης, κλήθη ο Πρόεδρος να δώσει γραπτή απάντηση επιστολή προς τον κύριο Μωρέρα ε, από τις μεταφορές ε, που θα κοινοποιηθεί φυσικά και στα μέλη. Επίσης, ε, ζητούμε από τους Επιτρόπους Κάλλας, Αρμούνια και Ντεγκούχη τα στοιχεία σχετικά με τον ανταγωνισμό στις μεταφορές. Να σχολιάσουν ιδιαίτερως την ε, ε, εξαγορά της UPS και της TNT. Επιτροπολογία. Οι συντονιστές ζήτησαν ε, από τον Πρόεδρο να ζητήσει από τον Επίτροπο Κάλλας ε, σχόλια για το καθεστώς το σχετικό με το υγραέριο και άλλα καύσιμα, ιδιαίτερα μετά την ε, χαλάρωση των μέτρων και της σχετικής απαγόρευσης, μετά στα υπόλοιπα θέματα, στα λοιπά, οι συντονιστές ζητούν από τον Πρόεδρο να συντάξει προφορική ερώτηση που θα συνοδευτεί από σχόλιο και απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη φορολόγηση των επιχειρήσεων σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη Γαλλία. Επιστολή επίσης του Προέδρου Μπαρόσο προς τον Πρόεδρο Σούλτς, για τα πολύ μεγάλα φορτηγά, τα λεγόμενα Megatrucks ε, και προ σωρινό χρονοδιάγραμμα. Που, θα, που αποφασίστηκε στη Συνεπιτροπή των Συντονιστών. Αυτά είναι όλα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν υπάρχουν σχόλια ως προς τις προτάσεις των συντονιστών. Σας ευχαριστώ θερμά. Και στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές TNT. με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, τον κύριο Κουμουτσάκο και τον κύριο Ερτού. Ερτού. Και ζητώ, με προτείνω μάλλον να δώσω το λόγο πρώτα στους δύο εισηγητάς και στη συνέχεια να ακούσουμε τον ε, κύριο Πάκε από την Οικονομική και Νοσηματική Επιτροπή. Ο καθένας από τέσσερα λεπτά Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Διορθώνων, κύριο Σπακ, και ε, στη συνέχεια να ακούσουμε ερωτήσεις και παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 4.30. Έχουμε περίπου μια ώρα στη θέσή μας και ως εκ τούτου ξεκινώ πρώτα με τον κύριο Κουμουτσάκο και μετά θα ακούσω τον κύριο Ερτού. Παρακαλώ κύριε Κουμουτσάκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να τονίσω την σοβαρότητα και την ιδιαίτερη σημασία που έχει το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορούν αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο αναπτυξιακό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 10-15 χρόνια, αλλά και μετά από αυτή την περίοδο. Σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία, σε μια εποχή που η ανάπτυξη και η μεγένθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει μεταβληθεί από στόχο σε πιεστική ανάγκη, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών έχουν αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Αυτό το υπογραμμίζω όχι μόνο εν ώψη της συζήτησης για τις κατευθυντήριες γραμμές που ξεκινάμε σήμερα, αλλά εν ώψη της μεγάλης συζήτησης για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, τα Multinational Financial Framework 2014-2020 και βεβαίως εν ώψη της συζήτησής μας σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής, σε δύο εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος, για το ΣΕΦ, για το Connecting Europe Facility. Αυτά τα δύο άλλωστε είναι στενά συνεδεμένα. Τώρα, Όσον αφορά ειδικά την έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές, θα ήθελα να αναφερθώ στις γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες που μας καθοδήγησαν τον συνάδελφο κ. Ερτούγκ και εμένα ως co-rapporteurs, ως συνσυντάκτες στην διαμόρφωση της πρότασής μας. Ο συνάδελφος κ. Ερτούκ θα αναφερθεί στα ειδικότερα σημεία των τροπολογιών που έχουμε καταθέσει επί της προτάσεως της Επιτροπής. Και οι δύο πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι μια στέρεη και καλή βάση, ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη συζήτησή μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις μας έχουμε συμβάλει στο να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της πρότασης Επιτροπής. Εκεί που κρίναμε, κάναμε την πρόταση αυτή πιο, ρεαλιστική και σε άλλα σημεία την κάναμε πιο φιλόδοξη πιστεύω ότι έχουμε πετύχει μια καλή ισορροπία. Έχουμε καταβάλει ειλικρινή προσπάθεια ώστε να ληφθούν υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανησυχίες και οι ευαισθησίες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πιστεύουμε ότι έχουμε εξαντλήσει σχεδόν τις δυνατότητες συμπερίληψης αυτών των ευαισθησιών στην πρότασή μας. Θεμελιώδης αρχή και κατεύθυνσή μας ήταν το εάν με τις προτάσεις μας εξυπηρετούμε την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία στο σχέδιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Πιστεύουμε ότι η λογική της νέας μεθοδολογίας των δύο επιπέδων, του κεντρικού δικτύου και του πλήρους δικτύου, καθώς και των διαδρόμων που ακολούθησε η Επιτροπή, επιτυγχάνει τρεις στόχους η νέα αυτή μεθοδολογία. Πρώτον, υπηρετεί και ενισχύει την αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Δεύτερον, οδηγεί στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ενσωματώνει ισοδυνάμως όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των μεταφορών στο πλαίσιο της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό, όπως ίσως έχετε δει στην πρότασή μας, έχουμε προχωρήσει μόνον σε πολύ περιορισμένης έκτασης και μικρής κλίμακας διορθώσεις και προσθήκες στους χάρτες, διορθώσεις και προσθήκες που βρίσκονται απολύτως, και θέλω να το τονίσω αυτό, μέσα στο πλαίσιο και σέβονται πλήρως την μεθοδολογία που έχει ακολουθεί από την Επιτροπή. Δεν τρέφω ψευδεστήσεις. Αντιλαμβάνομαι τον πειρασμό που υπάρχει σε πολλά μέλη της Επιτροπής, σε πολλούς συναδέλφους, να επιτύχουν κάτι καλύτερο όσον αφορά στη συμπερίληψη χωρών ή της περιοχής τους στους χάρτες και κυρίως στο κεντρικό δίκτυο. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω ταυτόχρονα να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Η αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και ο σεβασμός της μεθοδολογίας δεν είναι για μας διαπραγματεύσιμα. Αυτός ο κανονισμός δεν είναι τοπικού ενδιαφέροντος, είναι κανονισμός στρατηγικού χαρακτήρα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Όλοι θα πρέπει να θέλουμε ταχεία πρόοδο. Όλοι δεν θα πρέπει να θέλουμε να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και να μακρύνουμε αυτή τη συζήτηση σε σημείο που θα αντιστρέψει ή που θα καταστρέψει την προσπάθειά μας να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα παρακαλούσα επομένως τους συναδέλφους, με την βαθιά εκτίμηση και φιλία που τρέφω προς όλους, να λάβουν υπόψη τους αυτή τη βασική παραδοχή όταν θα ετοιμάζουν τις τροπολογίες τους. Προσβλέπουμε στην κατανόηση και στην καλή τους θέληση. Ως προς τα επιμέρους πεδία των αλλαγών που έχουμε κάνει, αυτά αφορούν κυρίως στην καλύτερη δομή και οργάνωση των στόχων και των προτεραιοτήτων, στην ενίσχυση της εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Θέλω να τονίσω ότι εδώ, στο σημείο αυτό, της ενίσχυσης της εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντολογικών ευαισθησιών, έχουμε αγγίξει τα όρια μας και το μήνυμα είναι ότι το περισσότερο δεν θα είναι κατά και καλύτερο. Το άλλο πεδίο είναι η αναγνώριση της μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην όλη διαδικασία των επιμέρους projects. Εδώ επίσης πιστεύω ότι έχουμε εξαντλήσει τις ρεαλιστικές δυνατότητές μας. Έχουμε κάνει επίσης αλλαγές όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό των διαφόρων projects. Επίσης, όσον αφορά την ενίσχυση της ενημέρωσης, της διαφάνειας και κατ' επέκταση της λογοδοσίας. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε ενισχύσει, πιστεύω, ουσιαστικά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το βασικό μήνυμα που πιστεύουμε και γι' αυτό θα μιλήσω στα αγγλικά, γιατί νομίζω ότι ενισχύεται η κατανόηση του μηνύματος. In the view of... Κατά την άποψη των εισηγητών, η πολιτική για την ευρωπαϊκή δίκτυο μεταφορών θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένη εν ώψη τη προσθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του στόχου του 2020, πιο συνεκτική και πιο συντονισμένη και πιο με περισσότερη διαφάνεια. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει η πολιτική αυτή να είναι πιο βιώσιμη, πιο αποτελεσματική, να βοηθάει τι νέε μεταφορέ για να αυθεντικό δίκτυο και αυθεντικά επίσης ευρωπαϊκή με μια σαφή ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Είμαστε ανοιχτοί και έτοιμοι να συζητήσουμε νέες καλές ιδέες και προτάσεις που θα κάνουν το χαρτί αυτό ακόμα καλύτερο. Και αυτό θα το κάνουμε σε στενή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και με τον καθέναν από εσά. Με τους σκιώδεις εισηγητές άλλωστε είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πριν από περίπου δύο μήνες στο Στρασβούργο. Αυτές είναι οι βασικές αρχές, οι βασικές σκέψεις που έχουν οδηγήσει την προσπάθειά μας, μια προσπάθεια πολύπλοκη και δύσκολη και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν γιατί είναι πολύπλοκη και γιατί είναι δύσκολη. Πιστεύουμε ότι έχουμε μπροστά μας και σας δίνουμε ένα ουσιαστικό, μια ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης της πρότασης Επιτροπής και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να το κάνουμε όλοι μαζί ακόμα καλύτερο. Όπως σας είπα πριν, ο συνάλφος κύριος Ερτούγκ με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολύ στενά και πολύ αποδοτικά πιστεύω αυτούς τους μήνες ε, θα ε, παρουσιάσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις προτάσεις που έχουμε εντάξει ε, στο χαρτί μας προσπαθώντας να κάνουμε καλύτερη την πρόταση της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σερτού. Αναλάβετε τη σκητάλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Κουμουτσάκος εξέθεσε τις κύριες αρχές που μας καθοδήγησαν στο έργο μας. Όντως, σημαντικό θεωρήσαμε και να συνεργαστούμε μαζί καλά και να επιτύχουμε τον, τον κύριο στόχο για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο των μεταφορών που κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του, που είναι ένα πραγματικό δίκτυο μεταφορών. Διαβάσαμε με ενδιαφέρον ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την θεωρούμε αρκετά καλή, όπως είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος, θεωρώ και εγώ ότι μπορέσαμε να τη βελτιώσουμε, να την εξειδικεύσουμε, να τη συγκεκριμενοποιήσουμε και εισάγοντας τους ε, ορισμούς να βοηθήσουμε και τον κάθε συνάδελφο ο οποίος δεν είναι εισηγητή, να αντιληφθεί γιατί πράγμα μιλάμε για το θέμα της χρηματοδότησης δεδομένης και της χρηματοοικονομικής ε, κρίσης ε, είχαμε μέχρι τώρα απουσία συντονισμού ως προς τα χρηματοοικονομικά μέσα και δεν μπορέσαμε και να ορίσουμε προτεραιότητες σε σχέση με την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Η διαφάνεια σημειώνεται επίσης στην οποία θέλουμε περισσότερες πρόοδους ε, που άλλωστε επιδιώκουμε πιστεύω και εξασφαλίζουμε με τις ε, τροπολογίες μας. Ο κύριος Κουμουτσάκος επίσης ανέφερε ότι εξ αρχής θεωρήσαμε και καλωσορίσαμε την πρόταση με τη μεθοδολογία που προτάθηκε και που μας επιτρέπει πιστεύω να έχουμε μία ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να άνοιγουμε τους ασκούς του αιώλου και να παραμένουμε και ακριβοδίκαιοι απέναντι σε κάθε περιοχή. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι περιφερειακά σχέδια ή έργα μπορεί να φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα ή γοητευτικά στον καθέναν, ναι, αλλά σας παρακαλώ αποφύγετε να κάνετε τέτοιε προτάσεις, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι διευρωπαϊκά δίκτυα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα συμβαστούμε σε ε, τοπικά σχέδια ή έργα. Αυτό που επιδιώξαμε εν γέννη να κάνουμε ήταν πρώτον ε, να επιτύχουμε τους στίχους του 2020, τα 2020 20 καλυτερα αλλά και τους στόχους ε, των περιφερειακών των, των αποτελεσματικών μεταφορών και θα ήθελα συγκεκριμένα να φέρω την οδηγία για την αποτελεσματικότητα των μεταφορών όπου απεδείχθη πολύ γρήγορα ότι δεν μπορούσαμε να επιτύχουμε το στόχο του 20%, μόνο το 10% μπορούμε να περιμένουμε ότι επιτύχουμε. Ε, και επίσης γνωρίζουμε όλοι ως ε, ειδικοί εδώ ότι υπάρχουν υπάρχει πρόβλημα ως προς τις εκπομπές του τοξιδίου του άνθρακα και αυτό ο τομέα των μεταφορών δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους όπως είχαν οριστεί στο, στην απόφαση 2020. Στους ορισμούς τώρα που συγκεκριμενοποιούμε. Συγκεκριμενοποιούμε τους ορισμούς Φερρυπίν, στο άρθρο 7, εκεί όπου γίνεται λόγος για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα και σαφώς σημειώνουμε ποια είναι αυτά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για μια κοινωνικο-οικονομική ανάλυση κόστους η οποία ισοδυναμεί με μια μικρή κλίμακα ε, impact assessment, μια αξιολόγηση κόστου αποτελέσματο, διότι θέλουμε, κυρίε και κύριοι συνέλφοι, να βλέπουμε τι επενδύσει στον χώρο των μεταφορών ω μακροπρόθεσμες φυσικά επενδύσεις σε όλες τις διαστάσεις των επιπτώσεών τους, θετικές ή αρνητικές. Γι' αυτό και θέλαμε αυτήν την κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση συνεπειών. Στο, στο άρθρο 4 επίσης ε, για τους στόχους. Στους στόχους ε, προβαίνουμε σε ένα σαφή ορισμό και πάλι έγινε λόγος για την ευρωπαϊκή προστέμενη αξία. Συχνά ακούμε να γίνεται λόγος για αυτήν και γι' αυτό θέλουμε πολύ συγκεκριμένα να διαπιστώνουμε ποια είναι αυτή η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ποια είναι λοιπόν είναι η προσθέμενη αξία ως προς την βίωσιμο, την αηφορία, ως προς την σύνοχη και ως προς την αποτελεσματικότητα αλλά και ως προς την βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της ωφέλειας, του ωφέλους που μπορούν να προσφέρουν τα έργα αυτά. Τέσσερις λοιπόν τομείς ε, που εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Προσθέμενη Αξία. Ω προς την χορύπαρξη επίση και ιδιαίτερα ε, στη σιδηροτροχιά, θέλουμε όχι μόνο να περιορίσουμε αλλά και να μειώσουμε την ε, ηχορύπανση Περιορισμός και μείωση λοιπόν της συγχωρήπανσης, ε, χωρίς, την οποία μείωση δεν μπορούμε να μιλούμε για συνοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική. Εδώ εξηγούμε και γιατί χρειάζονται οι επενδύσεις ως προς το τροχαίο υλικό, rolling stock, αλλά και γιατί σε περιοχές ε, όπου έχουμε μεγάλη πληθυσμιακή κάλυψη, Γερμανία, Γαλλία, αστικά κέντρα μεγάλα, ε, πρέπει να ικανοποιήσουμε και τις προσδοκίες των πολιτών για χαμηλά ποσοστά εκπομπής ε, ήχου, θορύβου. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά τις εσωτερικές πλωτές οδούς και που ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να δοθεί και από την σκοπιά των φυσικών πόρων και θησαυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλιστεί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι η χρυσή αυτή τομή, η βέλτιστη αυτή ισορροπία όπου με μία άριστη περιβαλλοντική νομοθεσία και άριστο επεδοτήρηση αυτή τη νομοθεσία μπορούμε και να αξιοποιήσουμε ως μέσα μεταφορά τι πλωτές οδούς μας. Αλλά πάντα σε σεβασμό με το περιβάλλον, αυτό το μεγάλο θησαυρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, για τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους, Motorways of the Serum, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να πω ότι δεν ήταν τόσο σαφείς οι προτάσεις και γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 να έχουμε σαφή εικόνα, σαφείς προτάσεις συγκεκριμένε για το πώς θα ενταχθεί και αυτή η πρόταση. Ο κύριος Κουμουτσάκος επίσης αναφέρθηκε στους ε, διαδρόμους corridors που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αποτελούν μέσα συντονισμού και υλοποίησης. Γιατί ήδη έχουμε μεν διαδρόμους, είναι γνωστό αυτό, αλλά θέλουμε αυτοί οι διάδρομοι, χωρίς βεβαίως να αποτελούν δεύτερες ή διπλές δομές, να αξιοποιούνται ως πραγματικοί διάδρομοι, ως μέσα δηλαδή για την επίτευξη των στόχων. Οι διάδρομοι θα ε, τελούν υπό τη διαχείριση ενός Ευρωπαίου ε, συντονιστή, θα καλύπτονται από μια Ευρωπαϊκή Συντονιστική Μονάδα. Όπως είπα υπάρχουν ήδη αυτοί οι διάδρομοι, αλλά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητούμε να υπάρχει μια ρητή αναφορά και στις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Συντονιστή της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Μονάδας ως προς τους διαδρόμους και ίσως και ενίσχυση ακόμη των σχετικών αρμοδιοτήτων. Επίσης, ο κύριος Κουμουτσάκος ανέφερε τη βασική αρχή της συμμετοχή της εμπλοκής στο εγχείρημα αυτό της τοπικής, του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου. Βεβαίως και θα πρέπει αυτό να επιτευχθεί η εμπλοκή, όπως είπα, του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου και θα εξασφαλιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η λήψη αποφάσεων σωστών όταν αυτός που λαμβάνει βαρύ συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος αυτός ο οποίος ε, είναι πιο κοντά στην υλοποίηση του έργου και όχι κάποιος ε, πολιτικός παράγων ή διοικητικός παράγων ο οποίος έχει μεγάλη απόσταση από το σημείο, από τον τόπο στον οποίο θα υλοποιηθεί το έργο. Γι' αυτό θέλουμε τοπικούς παράγοντες πάντα. Επίσης και κλείνοντας η υποχρέωση για λογοδοσία, ενημέρωση, διαφάνεια, η διαφάνεια και η ε, καταγραφή απολογισμών έχει πολύ μεγάλη σημασία όπως για κάθε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη καλούνται σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα και, για, και τις ε, απαιτήσει σε χρηματοοικονομικά μέσα να ενημερώνουν και να διαθέτουν στο το δυνατόν πιο λεπτομερή στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η ίδια υποχρέωση ενημέρωσης ε, υπάρχει και από πλευράς μας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι ποιε είναι οι δυνατότητε χρηματοδότηση. Είναι περίπλοκα τα χρηματοοικονομικά στην υπόθεση αυτή. Είναι αρκετά μεγάλο το πλέγμα και θέλουμε όσο το δυνατόν πιο ευρεία και διαφανή ε, εικόνα τη χρηματοοικονομική κατάστασης. Για να κλείσω θα έλεγα ότι είναι μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οποία είμαστε ευγνώμονε. είναι μια καλή πρόταση η οποία βελτιώνεται ωστόσο με τι δικές μας συγκεκριμένε προτάσει και παρακαλώ για άλλη μια φορά τις και του συναδέλφου, γιατί όλοι στο παρελθόν και ιδιαίτερα του τελευταίου τις τελευταίες εβδομάδες και μήνε ε, δραστηριοποιηθήκαμε στην υπόθεση αυτή και ασχοληθήκαμε. Οτιδήποτε ερώτημα έχετε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι ε, μην ε, διστάσετε να μας ε, το φέρετε να το συζητήσουμε, αλλά παρακαλώ οτιδήποτε πρόταση να μην περιέχει μόνο περιφερειακού ή τοπικού χαρακτήρα ε, ιδέες. Ας παραμένει το εγχείρημά μας αυτό ευρωπαϊκό. Και μια τελευταία παράκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δει τους εισηγητές, να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και δει τους εισηγητές για την εξέλιξη των ε, επαφών και των διαπραγματεύσεων με την ε, Κροατία, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ειδικά εμείς ποια είναι τα σχέδια, ποιο είναι το βασικό δίκτυο, ποιο είναι το, το κύριο δίκτυο ε, και αυτό πιστεύω έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενημερωθούμε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους σκιώδεις συγκητές για την πολύ καλή συνεργασία, την πολύ ειλικρινή συνεργασία που μας βοήθησε σημαντικά στο έργο μας. Είμαστε βέβαια στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Next, uh, Mr. Back from the Economic... τώρα από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχετε τέσσερα λεπτά κύριε Μπακ, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές στον κατάλογο. Tack så mycket, herr ordförande. Ehm, ja, några korta punkter om det eh, betänkandet. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα δευτερεύον σημείο να σας αναφέρω σε σχέση με την ε, γνωμοδότηση αυτή. Ο κύριος Μπακ. Εμείς στην Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή έχουμε εκπονήσει τη δική μας γνωμοδότηση όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των ε, δικτύων και η Επιτροπή μας ε, θεωρεί θετική και χαιρετίζει την πρόταση αυτή σε σχέση με τα δίκτυα αυτών των μεταφορών και συμφωνούμε για να υπάρχει αυτό το δίκτυο πυρήνα και το γενικό, το γενικό δίκτυο όπως επίσης και με τους διαδρόμους και όσον αφορά την Επιτροπή Μεταφορών εμείς θεωρούμε ότι οι διάδρομοι επίσης θα έπρεπε να υπάγονται ίσως αυτόν τον κανονισμό. Βεβαίως το θέμα εδώ είναι τι θα γίνει όσον αφορά την χρηματοδότηση. Και περιμένουμε πώς και πώς τις προτάσεις για την χρηματοδότηση εν του οργανισμού για το 2020 αλλά και για το 2030. Και θέλουμε τα σχετικά προγράμματα να ληφθούν υπόψη από το σχέδιο κανονισμού. Επίσης, θεωρούμε ότι μπορούμε περαιτέρω να βελτιώσουμε τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους αλλά και το δίκτυο πυρήνα και αυτό γιατί σε πάρα πολύ σημαντικές περιοχές όπως στην Βαλτική αλλά και στη Μεσόγειο έχουμε διασύνδεση σημείων. Επίσης είμαστε υπέρ βιώσιμων μεταφορών, καινοτομία και έτσι να έχουμε προσβασιμότητα σε εναλλακτικού τρόπους ε, καυσίμων. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο τους διαδρόμους. Θεωρούμε πάντως ότι αυτή η οδηγία είναι συνέχεια άλλων πρωτοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω η πράσινη διάδρομη. Και έχουμε επίση και άλλε πρωτοβουλίε οι οποίε ε, αξιοποιούνται σε διάφορα κράτη-μέλη και άρα και μπορούμε και εδώ να τις δανειστούμε. Συμφωνούμε επίση με την γνωμοδότηση τη δική σα ότι τα δίκτυα μεταφορών θα πρέπει να συγκροτηθούν με κριτήρια ουδέτερα. Και είναι σημαντικό το να μην έχουμε ρύθμιση υπερβολικά λεπτομερή στην οδηγία. Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικά εργαλεία πολιτικής και πάρα πολύ συχνά είναι δύσκολο να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα ε, του ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών. Μιλούμε για την προσθεμένη αξία την ευρωπαϊκή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουν πολλές φορές μονόπλευρη προσέγγιση όσον αφορά τις μελέτες επιπτώσεων. Έχουμε επίσης το πλήν 60% όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και μιλούμε επίσης για τις εκπομπές που προέρχονται από τα οχήματα και οι υπολογισμοί μας γίνονται από τη βάση αυτών και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ροή των, ε, της, της ε, κυκλοφορίας στο μέλλον. Να δούμε όμως τι είδους καύσιμα θα χρησιμοποιούν τα φορτηγά, τα γιοταχή, τα πλοία μέχρι το 2050. Νομίζω δε ότι θα ήταν αδύνατον να υπολογιστεί αυτό για οποιαδήποτε συγκεκριμένη επένδυση. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες για να έχουμε περισσότερη βιωσιμότητα. Έχουμε επίσης δύο βασικές κατευθυντήρες που είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά το πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το νομοθέτημα. Εμείς επίσης ε, ενδιαφερόμαστε για αυτό που διαφέρετε και εσείς γιατί θέλουμε να υπάρχει συνδιαχείριση των διαδρόμων και να μην κατησχίσουν τα εθνικά συμφέροντα και η ευρωπαϊκή προστιμένη αξία θα απειληθεί. Θέλουμε επομένω έτσι να γίνει διαχείριση και να μην υπάρξει υπερβάλλουσα γραφειοκρατία. Έχουμε μια αιτησία έκθεση όσον αφορά την ανάπτυξη των διαδρόμων, θέλουμε συγκεκριμένο μηχανισμό για αυτά τα προβλήματα και να μην υπάρχει έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι η συγκρότηση τέτοια υποδομής μεταφορών πολλές φορές προσκρούει στα τοπικά συμφέροντα. Όμως μπορούμε ε, με τον διάλογο με την τοπική κοινωνία να αποφύγουμε να μειώσουμε αυτά τα προβλήματα και έχουμε εμείς ε, ε, συντάξει έγγραφο για βελτίωση των διαβουλεύσεων όσον αφορά τα έργα υποδομής. Και σας ευχαριστώ που δώσατε το λόγο. Θα λάβουν τώρα το λόγο οι τρεις σκιώδες ηγητές. Mrs. Lichtenberger, Mr. Van Dalen, Mr. De Grandes, Mr. Ugias, and Mr. DeBacker. Is there anybody else wants to be added to that list? Mr. Grosch, and Mrs. Ayala, Mrs. Senalova because of course you are drastically now reducing your time each time. Προσοχή, μειώνεται τώρα το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Λέω ο πρόεδρος, καλώς. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Τρίλεπτο για τους και οδησηγητές και δίλεπτο για τους άλλους. Και το εννοώ, όχι δύο δέκα, δύο, δύο. Ξεκινούμε με την κυρία Μπιλμπά από τους φιλελευθέρους. Έχετε τρία λεπτά κυρία Μπιλμπά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους σας. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές γιατί πιστεύω ότι κάνανε εξαιρετική δουλειά δίνοντας ε, μεγαλύτερη σαφήνεια στο κείμενο της Κομισιόν και βελτιώνοντας το αισθητά. Τώρα, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να, να δούμε ξανά τον όρο προστιθέμενη αξία και την προστιθέμενη αξία που δίνουν τα έργα. Το θέμα της συμμετοχής ε, των πολιτών. Θα έπρεπε να καταβάλουμε μία προσπάθεια για να μπορέσουμε να στήσουμε καλά θεμέλια, να ανταλλάξουμε πληροφορίες, διότι έχουμε καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε, για παράδειγμα, τμήματα ε, ε, σιδηροτροχιών υψηλής ταχύτητας, τα οποία έχουν εκτελεστεί στην Ευρώπη, κατόπιν διαβούλευσης με τους ε, πολίτες. Επίσης το κόστος όφελος θα πρέπει και αυτό να το συμμεριστούμε με τους οφείλες, θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις μετά όχι μόνο τις κλιματικές αλλά και τις περιβαλλοντικές διότι έχουμε εμεί εμπειρία ότι πολλές φορές γραμμές υψηλών ταχυτήτων έχουν βαριές ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην αρχή της κατασκευής τους, αλλά μετά περιορίζουν την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με τα στοιχεία, ποιος είναι ο έλεγχος για να έχουμε έναν καλύτερο τρόπο ελέγχου και της βάσης αυτών των σχεδίων αλλά και του συστήματος χρηματοδότησης. Θα ήθελα να ενισχύσουμε, συμμερίζομαι δηλαδή αυτό που υπόθηκε και το λέω και στην Κομισιόν, για να μου πει τη γνώμη της. Να έχουμε λοιπόν έναν καλύτερο ορισμό για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας και να δούμε πώς τους ενσωματώνουμε στους στόχους. Γίνεται τώρα μια μικρή τροποποίηση μεθοδολογικού χαρακτήρα στην πρόταση της Κομισιόν. και κατά αυτόν τον τρόπο συμπεριλαμβάνονται η, η Κρήτη και τα Κανάρια νησιά. Σημερίζομαι αυτή τη γνω... την αλλαγή στη μεθοδολογία, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι λέει η Κομισιόν σχετικά με αυτό. Πάντως, ε, εγώ συμμερίζομαι σε πολλά από όσα λέγονται εδώ και θα καταθέσουμε και τις τροπολογίες που χρειάζεται για να δώσουμε παραπάνω προστιθέμενη αξία. Για τους πράσινους τρία λεπτά ο κύριος Κράμερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για μας είναι κάπως βελτιωμένη πρόταση. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια φυσικά και αυτό θα το επιτύχουμε χάρη στην, ε, στο, στην καταγραφή των λογαριασμών κτλ. Βεβαίω θέλουμε μια οικολογική διαμόρφωση των εσωτερικών πλωτών οδών, αλλά αυτό που έχουμε επικρίνει ανέκαθεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε να μην επιλύεται, δηλαδή το γεγονός ότι οι μεταφορές είναι ε, γεμάτο μπαλώματα, μια κουρελού γεμάτη μπαλώματα και δεν υπάρχει μια οργανωμένη δομή μεταφορών. Λείπουν από εδώ και από εκεί κάποια τούνελ ή στον άξονα Φερρυπίν Βαλτικής Αδριατικής λείπει το κόρα, λείπει το ζέμερι και κάποιες σύραγγες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί ε, αλλά δεν έχουν προχωρήσει. Από το Ζάγκρεπ στη Βιέννη ή αντίστροφα Βιέννη, Ζάγκρεπ, έξι ώρες μέσω της ε, κοιλάδας της Πανολικής χωρίς τούνελ, γιατί είναι μια εναλλακτική οδός. Όταν πρόκειται να φτιάξουμε σύραγγες, πρέπει να υπολογίζουμε διπλές λωρίδες, χρόνο, εργαλεία, σκάψιμο, κόστος μεγάλο και ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι πάντοτε αυτό είναι η καλύτερη λύση. Χαίρομαι επίσης ε, που υπόθηκε ότι θα πρέπει να εγκαταληφθεί ε, η λύση που, πάντοτε, που έχει μόνο περιφερειακό χαρακτήρα. Γιατί όμως εμφανίζεται σε φορές το Ηράκλειο ή γιατί η Λιέγη, η οποία είναι ένα αεροδρόμιο σε απόσταση μια ώρας από, την, ε, από τις Βρυξέλλες, εμφανίζεται τόσο πολύ μες στο σχέδιο. Γιατί να μην είναι το München Gladbach ή οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο. Το Στετίν του Βερολίνου, 30 χιλιόμετρα απόσταση και δεν έχει επαρκή ηλεκτροδότηση και άλλα αντίστοιχα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να, επικεντρωθούμε, να συγκεντρωθούμε στα ουσιαστικά. Παρίσι, Βρατισλάβα, το Ούλμα, όλα αυτά τα ζητήματα είναι, οι, οι διάδρομοι αυτοί είναι λύσεις καλές, ε, Ωστόσο, χρηματοδοτούνται με υπερβολικά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσω η προσθέμενη αξία ευρωπαϊκή να μην έχει εξασφαλιστεί πάντοτε σε όλε τι λύσει αυτέ. Άρα, θέλουμε τα 20. 30 χιλιόμετρα της παραμεθορίου που μπορεί να μην έχουν εθνική ε, σημασία και γι' αυτό δεν χρηματοδοτούνται από, τις, εθνικού τους αλλά έχουν τεράστια ευρωπαϊκή αξία να είναι αυτά στα οποία θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και να μην χρηματοδοτούνται Πλήρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη την έκταση τα σχέδια αυτά και οι διάδρομοι αυτή αλλά κυρίω οι παραμεθόροι περιοχέ. Ευχαριστώ πολύ, Τσίλερ Μισιάρ. Ε, και εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω του ε, συνεισηγητέ γιατί επένδυσαν πάρα πολλά, ασχολήθηκαν πάρα πολύ και επίσης ε, όλο το καλοκαίρι ασχολήθηκαν ε, με επιτυχία. για να δούμε τώρα μερικές διευκρινήσεις. Τι θα πει ε, στην, το 18 ο ορισμός της προστιμής αξίας. Νομίζω ότι εδώ βελτιώνουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης νομίζω ότι έτσι αυξάνονται οι ροές των μεταφορών μεταξύ των των μελών και νομίζω ότι το Συμβούλιο ε, δεν έχει αυτόν τον ορισμό και τέλος πάντων ε, έχει υιοθετήσει μόνο ένα τμήμα αυτού και ε, το θέμα είναι κατά πόσον έχουμε στα άρθρα 2, 8 και 4 τη σχετική μνήμα. Επίσης το 28 και το 24, αυτά τα δύο άρθρα ε, είναι όλα ορισμοί που δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζονται. Βέβαια καταλαβαίνω ότι έχουμε την τροπολογία 29 όσον αφορά του, τις τέσσερις κατηγορίες των στόχων, αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα, κάλυψη όλων των ε, επιλεξίμων και χρηστών και συνοχή. Ωραία όλα αυτά, όμως από την άλλη μεριά συμφωνώ με αυτό το οποίο προλίγο ο κύριος Κράμερ, ότι δηλαδή ε, στις περιφερειακές ε, ε, χώρες ή στις περιφέρειες των άκρων της Ένωσης έχουμε κάποιο είδους αποκοπή από το κέντρο για ιστορικούς λόγους και νομίζω ότι τελικά δεν είναι θέμα μόνο των φραγμών των γεωγραφικών αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε και τους πολιτικούς φραγμούς και εμπόδια. Παρακάτω τώρα όσον αφορά τα κριτήρια τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα. Εγώ ε, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που οι συντάκτες του κειμένου ετήρησαν ε, την προσέγγιση στο 57, στο 60 και στο 61 μέχρι 63, την προσέγγιση κατά διάδρομο. Ε, νομίζω ότι το Συμβούλιο δεν έχει πρόθεση να διαγράψει, να μην ακολουθήσει την προσέγγιση των ε, ε, διαδρόμων και έτσι να συρρυκνώσει την προσθέμενη αξία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι η καρδιά της πρότασης και αυτό πρόκειται να ισχύσει την επόμενη πταετία. Και επίσης εγώ θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να την υπόψη ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προσέγγιση αυτή. Ε, επίσης θα πρέπει τα προγράμματα ε, των διαδρόμων έχουν προτεραιότητα σε σχέση με, τη, με, τα έργα του πυρήνα. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Φρικέ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα εκφραστώ ως συνεισηγητής με την Ινές για τον ε, μηχανισμό του ΣΥΡ να συγχαρώ τους εισηγητές για τη δουλειά τους και να του συγχαρώ επίσης γιατί συνεργάστηκαν μαζί μας, κάνανε όλη τη δουλειά μαζί μας. Ε, γιατί ήταν δύο κομμάτια του ίδιου μηχανισμού και είχαμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Σημερίζομαι τις απόψεις για τη μέθοδο και παρακαλώ τον ε, Γιώργο να μου δώσει γραπτός αυτά τα οποία είπε. εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, λιτότητα, την αυστηρότητα του να μην παραμένει κανείς ε, στα κριτήρια τα οποία δόθηκαν επίσης ε, στο γεγονός ότι είναι βανάγνωστη η έκθεση διότι εδώ πρόκειται για ένα τεράστιο και πολύπλοκο μετανο. Εγώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πρέπει να πω ότι οι μελέτες εκ των προτέρων, οι εξάντε μελέτες με πολλαπλά κριτήρια είναι σημαντικές, δεν πρέπει να επιβαρυνθούν, δεν πρέπει να καθυστερούν, πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία. Ε, δεν θα πρέπει όμως να είναι κάτι το οποίο να βουλιάζει τα σχέδια και αυτό λόγω του βάρους της διαδικασίας. Ε, θέλω να πω ότι η έκθεση που μας παρουσιάστηκε είναι εξαιρετική. Αποτελεί Εδώ έχουμε ε, το, όχημα. Μετά χρειάζεται να βάλουμε τη μίζα και τη μηχανή για να ξεκινήσει αυτό το όχημα. Δεν πρέπει λοιπόν να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα αυτή την έκθεση, θα πρέπει να την αφήσουμε λειτουργική όπως είναι. Ο κύριος Αλχαδράουη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τους εισηγητές για την καταπληκτική τους δουλειά ουσιαστικά υποστηρίζουν τη θέση την αφετηρία της Κομισιόν. Εμείς ως Κοινοβούλιο πάντοτε είχαμε αυτή τη θέση. Είναι πολύ σημαντικό εμείς να κρατιόμαστε πάντα σε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία για να υποστηρίξουμε με μονομένα σχέδια τα οποία υποστηρίζουν αντικειμενικά σχέδια και με, συγκεκριμένους, με συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου, δηλαδή διασυνοριακή συνεργασία κλπ. Επίσης μεγάλη τεχνική διαλειτουργικότητα που θα πρέπει να, να είναι εγγυημένη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκαθαρίζουμε εδώ ορισμένου στόχους, δηλαδή τοπικές κοινωνίες οι οποίες συμμετέχουν πιο άμεσα, Τώρα εμείς ε, θα έχουμε ε, τίποτα ε, ψηλοδιορθώσεις να κάνουμε όσον αφορά στις ε, επιπτώσεις. Ε, για παράδειγμα έχουμε την τροπολογία 44 που αφορά στο Natura 2000 και τους, ε, τις περιοχές που βγαίνουν από το πακέτο άλλες φορές δικαιολογημένα, άλλες αδικαιολόγητα. Πρόκειται πάντως για ένα κείμενο, ένα κείμενο βάσης που μπορούμε να συνεχίσουμε. Μάλιστα για δύο λεπτά. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστώ πολύ τους ε, δύο εισηγητές για τη δουλειά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε του ασκού του αιώλου. Δεν πρέπει. Πρέπει να αποφύγουμε να ανοίξουμε του ασκού του αιώλου και να, για αντιθέτω πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα τα σημαντικά, εκεί που έχουμε τις, ε, τα, τα κύρια ζητήματα, εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα. Στη δική μου την περιοχή λοιπόν ε, και ξέρω ότι διαγράφει η πρόταση που αφορούσε τη δική μας ε, περιφέρεια και το, τους ε, υδάτινους δρόμους, από το Συμβούλιο μάλλον, ε, θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσε ίσως να εξεταστεί για ποιο λόγο διαγράφει αυτή η πρόταση το έργο και αν υπάρχουν και αντίστοιχα άλλα παραδείγματα. Ευχαριστώ κύριε Λίκτινμπέργκερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να απευθύνω εκ μέρους και του συναδέλφου βεβαίω Κράμερ, ο οποίο ε, βιάστηκε ε, να μιλήσει. Ε, θα ήθελα να εκφράσω λοιπόν τι ευχαριστίε μου προ του δύο συναδέλφου και θα προσπαθήσω χωρί να είμαι ηρωνική ή κοινική να πω ότι βλέπω με ενδιαφέρον ένα σχέδιο φιλόδοξο το οποίο όμως ε, σε τελικό αποτέλεσμα παραμένει στα ιωθώτα και σε μια προσπάθεια να διαφυλαχθούν ε, κάποια εθνικού επίπεδου ε, κέρδη ή ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να κοιτάξουμε σε περιπτώσεις όπου ένα κράτος βρίσκεται σε, μια, σε ένα αδιέξοδο με την έννοια ότι Φερρυπίν ε, λόγω μεγάλων χρεών δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιων έργων. Ε, θα ήταν μάλλον αυταπάτητο να λέμε ότι το αφήνουμε ε, και ξαναρχόμαστε σε πέντε χρόνια να κοιτάξουμε τι έχει προκύψει. Επίσης, όταν ε, λέτε ότι θα επαληθεύουμε, πότε είναι το ερώτημα, πότε θα επαληθεύεται η αξιοποίηση των κονδυλίων. Θέλουμε λοιπόν να βλέπουμε ξεκάθαρα την ε, αξιοποίηση και τα ωφέλη από την αξιοποίηση των πόρων. Στη συγχρηματοδότηση όταν δεν είναι δυνατόν να την προσφέρει ένα κράτος μέλος λόγω οικονομικών πιέσεων, δεν θα πρέπει αυτό κάπου να καταγράφεται για να μην χάσουμε και την αξιοπιστία μας. Για τη τελευταία ανάλυση και θέση εργασίας και Και μην ξεχνάμε ότι εδώ πρόκειται για οχταπλάσιες θέσεις εργασίας σε σχέση με την, όταν έχουμε να κάνουμε κατασκευή επίγειων δομών σε σχέση με τις υπόγειες δομές, οχταπλάσεις τις εργασίες ε, ας μην χάσουμε λοιπόν την αξιοπιστία μας. Λυπάμαι. Λυπούμε που μετά από τόσους επένους προς τους εισηγητές, εγώ θα διακόψω αυτήν την ε, σειρά επένων. Εγώ απαγοητεύτηκα. Είχαμε μία πρόταση της Κομισιόν και τη χειροτέρεψαν σε τρεις άξονες τις ε, ε, ναυτιλιακές ε, οδούς που επίσης τις πνίγουν με την τροπολογία 44 η οποία συσσωρεύει ένα σωρό αιτήματα Δηλαδή ε, δεν μπορούμε εμείς ε, να, να, να, να ξεκολλήσουμε ούτε ένα φύκι όταν φτιάχνουμε αυτές τις ναυτιλιακές οδούς. Μα εδώ υπερβάλλουμε. Και στρεβλώνεται και ο ανταγωνισμός. Δεν ξέρω, αυτή την τροπολογία τώρα τι να πω. Μπορεί να την ετοίμασε ο Κράμερ στο γραφείο του υπέρ της μπουντες των γερμανικών σιδηροδρόμων... και των σιδηροδρόμων γενικά. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Εδώ πρέπει να αφήσουμε τις εθνικές αρχές με την ησυχία τους έχουν τη δική τους άποψη. Αν μπούμε σε λεπτομέρειες δηλαδή, στην Ολλανδία δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ακολουθήσουμε τις δικές μας διαδικασίες, οι οποίες είναι μια χαρά. Η ανάλυση κοινωνικού κόστους ωφέλους, άμα θέλετε να μπλοκάρετε κάτι, μα αυτή την ανάλυση ξεκινήστε με το κοινωνικό-οικονομικό κόστος και, και το όφελος. Μετά έχουμε και άλλες ε, περίεργες προτάσεις αεροδρόμιο του Κάλιαρη και διάφορα τέτοια. Εγώ σέβομαι όλη αυτή την πολλοπλασιαστική τάση, αλλά εγώ θα θέσω φραγμούς με τροπολογίες. Ο κύριος Δεγκράντες. Ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη μας η μεθοδολογία που ε, θέτει η Κομισιόν είναι πολύ λογική και οι εισηγητές την εφαρμόζουν πολύ σωστά. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί η Κομισιόν ε, αφήνουν ε, έξω ορισμένε εθνικές ε, εμπνεύσεις αλλά εντάσσει άλλες. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Εμείς θα κάνουμε τροπολογίες που ίσως θα αφορούν εθνικά σχέδια μεν, αλλά θα είναι κοινού συμφέροντος με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Με το λιμάνι του Βίγκο στην Γαλλικία που είναι το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι στην Ευρώπη που δεν συμπεριλαμβάνεται. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρει η Κομισιόν που αφορά ε, στο τούνελ των Πυρηναίων μεταξύ Γαλλίας ε, και Ισπανίας που ακόμη εκκρεμεί. Θα πρέπει να ενισχύσουμε εμεί τους δρόμους για τα επόμενα χρόνια για περιβαλλοντικούς λόγους. Σύμφωνοι η έκθεση, είναι μια ρεαλιστική έκθεση. Εξετάζει την, τα θέματα οικονομικής συνοχής, ε, παίρνει τις ορεινές περιοχές υπόψη, τα νησιά και όλες τους τις ιδιομορφίες όπως και τις ιδιομορφίες των κρατών μελών τις οποίες ε, αφορούν αυτές οι διασυνοριακές συνδέσεις. Τώρα, είναι μια λυπητερή ιστορία η ιστορία αυτής της υπόθεσης. Είχαμε πρώτα 20 δις, μετά γίνανε 8 και άρχισαν και οι εκπτώσεις. Λοιπόν, μην μπούμε πάλι στις εκπτώσεις και έτσι πεθάνει ένα όνειρο. Ευχαριστώ πρόεδρε Σίμψον, λέει ο κ. Ζούτζες. Εγώ θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου στους δύο εισηγητές και στον κύριο Κουμουτσάκο και στον κύριο Ερτού. Κάνανε εξαιρετική δουλειά. Και πιστεύω ότι ξεπέρασαν αυτά τα όρια τα οποία έθετε η πρόταση της Κομισιόν. Και το κάνανε όχι βάζοντας τελίτσες πάνω σε ένα χάρτη, αλλά κρατώντας σταθερά τα κριτήριά τους. Δηλαδή, ορίζουν τις αρχές που διέπουν αυτήν την ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι στόχοι 2020 που πρέπει να μείνουν αμετάκλητοι όπως και τα άλλα κριτήρια τα οποία απαιτούν κοινωνικο-οικονομική ανάλυση ούτως ώστε αυτή η προπτική να αποκτήσει την προστιθέμενη αξία που καθορίζεται από τον προγραμματισμό. Θέλω τώρα εδώ να επικαλεστώ μια ειδική πτυχή, πέρα από το γενικό δηλαδή, διότι μέχρι τώρα οι, οι εισηγητές θησάβρισαν ότι ε, από τις, ε, τον καρπό των συζητήσεων είχαμε εμείς ε, στο, στην ακρόαση του Μαΐου ένα πρόβλημα με το θέμα των νησιωτικών περιοχών όπου κόπηκαν εντελώς ε, νησιωτικές περιοχές με εκατομμύρια κατοίκους ε, στην Μεσόγειο και εκτιμώ ιδιαίτερα εγώ τις τροπολογίες που έγιναν για να συμπεριληφθεί η Σαρδινία, η Κρήτη και όλες εκείνες οι προσδοκίες για οικονομική ολοκλήρωση, ολοκλήρωση ούτως ώστε να υπάρξει ομοιογενής ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Γκος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα εν συντομία να πω ότι αυτή τη φορά η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι καλύτερη ότι έχουμε δει στο θέμα αυτό και ως προς το πνεύμα και ως προς τη μέθοδο που έχει επιλογή. Ξέρουμε ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι αυτό το θέμα των μεταφορών είναι ένα σύνολο και δεν πρέπει να χαθούμε μέσα στις λεπτομέρειες. Εδώ ξέρουμε ότι μπορούν να αποδώσουν τα έργα όταν υπάρχει και η κατάλληλη χρηματοδότηση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα θέμα αργότερα σήμερα για το θέμα της χρηματοδότησης, το ξαναδούμε. Διαφάνεια. Και εδώ θα ήθελα να φερθώ σε κάποιες πτυχές ε, από μελέτες ε, που αφορούν προηγούμενες εμπειρίες και οι οποίες επισημαίνουν τον κίνδυνο το 80% των, της χρηματοδότησης να το απορροφήσουν μελέτες και μόνο 20% να μείνει για τα έργα στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη και βεβαίως όταν μιλούμε για την προσέγγιση της φύσης πρέπει να την ε, δούμε με σοβαρότητα, πρέπει να την επιδιώξουμε χωρίς ωστόσο να χάσουμε και την ουσία της υλοποίηση των έργων των μεταφορών. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω ότι η λύση η σχετική με την ε, παρουσία των κρατών όπως θα προχωρήσει εν τέλει θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή πρέπει βεβαίως να υπάρχει κεντρική ε, θεώρηση πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και τα κράτη-μέλη, το καθένα από πλευρά του, να κάνει τη δουλειά του, να υλοποιήσει το καθήκον που αναλαμβάνει ε, και να μην γυρίσει ο καθένας στη γωνιά του αγνοώντας ε, τις συμφωνίες και τα σχέδια που θα έχουν ε, οριστεί. Ελπίζω ότι θα καθένα θα μπορέσει να συμβάλλει δηλαδή από πλευρά του στην πρόοδο αυτού του εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστίες προ τον κύριο Αρτού και στον κύριο Κουμουτσάκο για το έργο το οποίο επετέλεσαν και για την ανάλυση τη μεθοδολογία αλλά και ε, τα όσα έχουν αναφέρει εδώ. Ε, ναι, και εγώ θεωρώ, όπως είπατε, να γίνει διάλογος για να αναθεωρήσουμε την μεθοδολογία. Είναι λογικά αυτά που προτάθηκαν για να, να άρουμε κάποιες παραλήψεις, κάποια λάθη, κάποιες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν να κάνουμε ε, στην Λασπάλμα, στην Κραν Κανάρια, εκεί για παράδειγμα, εκεί θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τι ισχύει εκεί για τη σύνδεση με την ε, Τενερίφη, μπορεί εκεί επιφέρει να γίνει μια τροπολογία και έτσι και η Τενερίφη να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το σύστημα επίσης. Φυσικά και συμφωνώ με όσα είπατε για το Βίγο και οπότε φυσικά και υπάρχουν κάποια κενά. Ε, αυτά πρέπει να τα δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε τους εμπειρογνώμονες, από τα κρατή-μέλη που ασχολούνται με αυτά και... Ε, όμως κάποιοι, τι, τι έγινε, κάποιες ρυθμίσεις εξαφανίστηκαν όπως το κανάλι του Λίμπεκ, στα Πυρηναία, Αλχεσίρας. Ε, αυτή είναι αυτός ο διάδρομος που ενώνει νότο προς με βορρά. Εξαφανίστηκε όμως, οπότε για όλα αυτά τα ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα ε, θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα γίνει ούτως ώστε να μην χαθεί η ουσία αυτού, του, του οράματος που είναι πάρα πολύ ευρωπαϊκό ε, για λόγους ε, καθαρά εθνικής ε, επικουρικότητας και επίσης από την άλλη μεριά λόγω της οικονομικής κρίσης είπαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι κατάχρεωμένα τα κράτη-μέλη, όπως ακόμα και η Γερμανία που χρωστά περισσότερο από την Ισπανία όσο και αυτό το παράδειξο. Όμως η Ευρώπη, η Ευρώπη δεν είναι κατάχρεως ε, επομένως, ο δρόμος που ακολουθήσουμε θα είναι τα ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα για να βοηθήσουν την οικονομία την ευρωπαϊκή. Όπως θα είπε ο κύριος Γκρός, ε, θα πρέπει και οι τομείς και επιμέρους να θεωρηθούν ως ε, συγκινούντα δοχεία. Ευχαριστούμε κύριε Κομισιόν. Λαμβάνει πως θα πει και Θα πρέπει να συζητήσουμε από κοινού αυτούς τους δύο κανονισμούς και να δούμε τι θα γίνει με την τροπολογία 57 η οποία ε, είπε ότι η προβλέπει να, την, την από κοινού εξέταση των παραρτημάτων. Την ε. Ευχαριστώ τους ηγητές, αλλά επίσης έχω και Κάποιε παρατηρήσει Συμφωνώ με τον κύριο Βαντάλεν και για την τροπολογία 44, η οποία θεωρώ ότι δεν στέκει εκεί που πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και κατασκευής έργων υποδομής. Για τις περιφερειακές αρχές νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εμπλακούν. Αρκούν οι εθνικές αρχές και ε, να γίνει στα πλαίσια εκείνα η διαβούλευση για να μην κολλήσουμε και μετά δεν γίνεται αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν αναφέρονται οι εσωτερικές πλωτές οδοί και τα σχετικοί λιμένες, όλο γιατί με τη θάλασσα ασχολούμαστε. Άρα θα πρέπει και εκεί να δούμε ποιους λιμένες θα συμπεριλάβουμε. Όσον αφορά τον σιδηροδρόμους, ε, το TSI και την διαλειτουργικότητα και είπαμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί το ζήτημα. Η διάδρομη είναι μια καλή ιδέα, όμως θα πρέπει οι ρυθμίσεις να είναι σαφείς και να μην έχουμε μεγάλο διοικητικό βάρος και γραφειοκρατία. Τα δίκτυα των μεταφορών θα λειτουργήσουν μόνο εάν η πρικοδότηση είναι επαρκής και γι' αυτό και θέλω να ζητηθεί από τα κρατη να διαθέσουν αρκετούς πόρους. Και θα μπορούσαν να ελκύσουν ε, επειδή τομέα, θα μπορούσαν ε, να εκδώσουν κάποια ομόλογα για τα έργα. Υπάρχουν ένα σωρό εναλλακτικέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τους δύο και εισηγητέ για την έκθεση, η οποία βελτιώνει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαντικά. Οι συνεισηγητές καθιστούν πιο συγκεκριμένο το κείμενο, ενισχύουν όρους όπως η ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία, τα κριτήρια αξιολόγησης ε, των έργων δημοσίου συμφέροντος, η αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, ε, η διασύνδεση ως προς τη Λευκή Βιβλό για τις μεταφορές έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Ίσως θα έπρεπε ωστόσο να υπογραμμίσουμε περισσότερο ότι χρειάζεται περισσότερη συνοχή κοινωνικο-οικονομική, αλλά και εδαφική συνοχή. και θα ήθελα να δω περισσότερε τροπολογίε στο θέμα αυτό τη εδαφική συνοχή. Ε, βέβαια, ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και η υλοποίηση των στόχων, ε, αλλά αυτά ήδη τα, τα ανέφεραν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τιτσά. Πρόεδρε, θα, θα αρχίσω με παρατηρήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία. Για την τροπολογία 11 οι δύο οι εισηγητές θέλουν να βελτιώσουν την μεθοδολογία της ε, Κόμισιον. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση η Κομισιόν να ορίσει μια μεθοδολογία που θα την έχουμε ως παράρτημα του κανονισμού. Δεύτερη παρατήρηση. Η εσωτερική, ε, τα εσωτερικά ε, λιμάνια θα πρέπει ε, να τα έχουμε Αυτά τα εσωτερικά λοιπόν πλωτά λιμάνια να τα έχουμε στην, σε ένα παρονισμό. Επίσης εγώ καταθέτω τροπολογίες όπου λέω ότι θα πρέπει ως αστική ε, ε, κόμβη να μπουν οι κόμβοι της Βραήλας και το λιμάνι επίσης ο κόμβος μεταξύ Γαλατσίου Βραήλας. Επίσης ε, μιλάμε και για την προτεραιότητα των πολυσυνδυασμένων μεταφορών. Να έχουμε έναν καλό συνδυασμό μεταξύ των εσωτερικών ε, ο, λιμανιών και των αυτοκινητοδρόμων. Διότι αυτά τα λιμάνια δεν τα έχουμε σήμερα ε, στην πρόταση της ε, Κομισιόν. Τώρα υπάρχουν και χώρες που έχουν μεγάλα σύνορα ε, δεν θα πρέπει με τους, ε, με τους γείτονές τους, δεν θα πρέπει να έχουν μόνο ένα ε, συνοριακό πόρεσμα, θα πρέπει να έχουμε πολλά περάσματα και θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Κύριος Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε κι εσείς να τηρήσετε το χρονικό όριο, κύριε. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα πάντως θα σας δώσουν πέντε λόγια για να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα τηρηθεί το όριο. Κύριε Πρόεδρε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όπως και οι βουλευτές θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η έκθεση και κινείται στο πνεύμα της δικής μας προτάσεως ε, η οποία παρουσιάζει αυτό το δίκτυο των μεταφορών το ευρωπαϊκό, το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό και πιο βιώσιμο και επίσης θα δίνει ένα βιώσιμο πλαίσιο για έργα υποδομής και πολιτικές, ούτως ώστε αυτές να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή πολιτική. βαστούμε τους συζητητές για το κείμενο. Ε, υπάρχει βελτίωση, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να βελτιωθούν περισσότερο Έχουμε ακόμα κάποια θέματα διατύπωση, θα συζητούμε με του συζητητέ και κυρίω όσον αφορά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ε, τι επιπτώσει στο εναλλαγή του κλίματο, στο CDA και θα πρέπει να χτενίσουμε την, ε, το κείμενο για τη διατύπωση για να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει και επίσης όσον αφορά τις διοικητικές επιπτώσεις θα πρέπει να το συζητήσουμε για να το αναλύσουμε. Έχουμε επίση δύο τροπολογίε που έχουν καταθέσει διάφοροι βουλευτέ για πώ μα προβληματίζουν. Η πρώτη είναι η αναθεώρηση που είπατε να γίνει όσον αυτό τι ισχύει για τους αυτοκινητοδρόμου του θαλάσσιους και εδώ υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του ότι θέλουμε να, τι θέλουμε να γίνει το 2013 και μετά μέχρι το 2013 λέει να γίνουν ε, να γίνει η αναθεώρηση, όμως τέλος πάντων έχουμε συμφωνήσει ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση και πιστεύω θα συμβαίνει με τους ηγητές. Το 44. Συμφωνούμε. Ποιος θα γίνει το δρόμο, ότι θα πρέπει ε, οι περιβαλλοντικές διατάξεις να εφαρμοστούν και επίσης ε, είπαμε ότι αυτό θα ισχύει για όλους τους τομείς όπως και το κείμενο που υπήρχε για το 1944 προβλέπει συμμόρφωση με τις ε, φιλοπεριβαλλοντικές διατάξεις και επειδή θα πρέπει να εφαρμοστούν στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου. Επομένως, θα πρέπει με τους ε, συνεισηγητές να δούμε ότι καλύπτονται οι στόχοι μας, αλλά θα πρέπει να τηρηθεί και η απαγόρευση του χώρου στις εσωτερικές πλωτές Τώρα, σαν την ουσία της ε, έκθεσης, έχουμε δύο σημεία. Έχουμε εντυπωσιαστεί ε, από το κείμενό σας. Ας πρώτα-πρώτα πρόκειται για τους ε, διαδρόμους. Νομίζω ότι το κείμενο είναι πιο συγκεκριμένο, πιο λειτουργικό και διευρύνει αυτούς που θα εμπλακούν τοπικούς παράγοντες περιφερειακούς. Άρα εδώ ε, παίρνει άριστα η θεώρηση του κειμένου μας. Μεθοδολογία. Χρησιμοποίησαν οι τη μεθοδολογία μας, ακρόαση και με συνέπεια κάνατε ό,τι και εμείς, κάνατε πάρα πολύ λίγες ε, τροπολογίες. Άρα το γράμμα και το πνεύμα της μεθοδολογίας μας το έχετε δανειστεί και με ανακούφιση συνειδητοποιώ ότι θέλετε να συνεχίσετε σε αυτό το πνεύμα. Θα βελτιωθούν οι χάρτες, αλλά αυτά τα δίκτυα που προβλέπονται θα συνεχιστούν και θα αναπτυχθούν μέχρι το 2030 και θα έχουν μια στέρεα πολιτική ω θεμέλιο. Σε ευχαριστώ κύριε Κομοτσάκο, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε <clears throat> και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερω όλου του συνάδελφου που συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση και εκείνους που αντιμετώπισαν θετικά την προσπάθειά μας αλλά και εκείνους και θα έλεγα περισσότερο εκείνους που άσκησαν κριτική. Διότι υπάρχουν επιχειρήματα που θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. Τώρα, όσον αφορά στα επιμέρους ζητήματα που θύχθηκαν, επιγραμματικά θα πω. Πρώτον, όσον αφορά, ε, και ξεκινάω γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, την χρηματοδότηση του project και την ε, δυνατότητα που υπάρχει από τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν οι μη. Κοιτάξτε, εμείς εδώ παρουσιάζουμε το σκελετό του αυτοκινήτου. Αυτό το αυτοκίνητο όσο καλά και αν είναι δομημένο, δεν μπορεί να κινηθεί αν δεν έχει μια αντίστοιχη ποιότητα μηχανή. Και αυτό είναι η χρηματοδότηση. Όλοι ξέρουμε ότι σε αυτό υπάρχουν δύο μεγάλες εκκρεμότητες. Η συζήτηση για, τις, για τον προπολογισμό 14-20 και η συζήτηση για το, για το Connecting Europe Facility, για το ΣΕΦ. Επίσης, συνδέεται με αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα των project Bones, των ομολόγων έργου. Εκεί, όπως γνωρίζετε, όλοι έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή, ειδικά ο συνάδελφος κύριος Κάνσιαν δίνει ένα πραγματικό αγώνα για να έχουμε μια βελτίωση. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι η συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τα guidelines. Αναγνωρίζω απολύτως την σοβαρότητά της, αλλά εκφεύγει, αν θέλετε, του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Όσον αφορά ε, τα υπόλοιπα που ακούστηκαν. Γιατί προσθέσαμε ε, νέους ορισμούς το κάναμε με έναν μόνο σκοπό. Όλοι οι συνάδελφοι, όλοι που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια να έχουν μια γενική εικόνα για το τι μιλάμε, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες παρανόησης για βασικές έννοιες όπως η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία ή η διαλειτουργικότητα κλπ. Ελπίζω η προσπάθειά μας αυτή να έχει βοηθήσει στο να γίνει πιο σαφές το κείμενο. Όσον αφορά ε, την συζήτηση για τα Motorways of the Seas, άκουσα και με προσοχή την ε, παρατήρηση της Επιτροπής, ε, δεν μπορεί σε ένα τέτοιο μεγάλο project που αφορά όλους τους τρόπους μεταφορών, η θαλάσσια διάσταση να είναι υποβαθμισμένη. Ο σκοπός λοιπόν της τροπολογίας μας, που μπορούμε βεβαίως να συζητήσουμε, είναι να μην είναι υποβαθμισμένη η θαλάσσια μεταφορά που είναι και φιλική προς το περιβάλλον και που μπορεί να γίνει φιλικότερη αναφυσβήτητα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών και πώς το βλέπουμε. Εμείς έχουμε ένα σκοπό. Όχι να εμποδίσουμε την υλοποίηση των projects, αλλά να τη διευκολύνουμε. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο όταν ξεκινά η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου σχεδίου να σταματήσει και τότε να λύνουν τα προβλήματα από το να έχει υπάρξει από την αρχή μια κατανόηση και συμφωνία όλων των παικτών, ώστε όταν ξεκινήσει το σχέδιο να υπάρχει βεβαιότητα και στις αγορές, αλλά και σε αυτούς που επενδύουν, ότι το, σχέδιο θα προχωρήσει. Αυτή λοιπόν ήταν η λογική, να, να βοηθήσουμε και όχι να εμποδίσουμε. Κρατάω τελευταίο και θα μείνω σε αυτό, το θέμα της μεθοδολογίας. δεν την ακολουθήσαμε τυφλά και ως λευκή επιταγή την μεθοδολογία που πρότεινε η Επιτροπή. Γι' αυτό το λόγο διοργανώσαμε μεγάλο, μια μεγάλη εξαντλητική δημόσια συζήτηση, ένα public hearing. Και από αυτό προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα σεβαστήκαμε, γι' αυτό είναι πολύ περιορισμένες οι τροπολογίες, σέβονται απολύτως τη λογική της μεθοδολογίας και είναι μέσα στο πλαίσιό της. Δεν εξυπηρετούνται παρά το γεγονός και το λέω παρά το γεγονό ότι στη συγκεκριμένη πρόταση υπάρχει το λιμάνι του Ηρακλείου πρέπει να σα πω ότι αυτό δεν προέκυψε επειδή τυχαίνει ο ένα εισηγητή να είναι Έλληνα, αλλά επειδή προέκυψε από τη δημόσια συζήτηση και δεν το έθεσε Έλληνα, αλλά γιατί ήταν μια μεγάλη συζήτηση που έκανε αυτέ τι διορθώσει. Εάν υπάρξουν και άλλε τροπολογίε, οι οποίε όμω σέβονται απολύτω τη λογική τη μεθοδολογία και δεν δημιουργούν προποθέσει ανατροπή τη, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Τελευταίο, το θέμα της Κροατίας πρέπει να μας απασχολήσει, διότι η Κροατία γίνεται σύντομα πλήρες μέλος, επομένως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, και αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε με την Επιτροπή, ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, μια, μια, μια, ένα de flexibility, αν θέλετε, στην, στο, ώστε να ληφθεί το θέμα της Κροατίας υπόψη, εάν βεβαίως πάμε σε πρώτη ανάγνωση, έτσι, γιατί αν πάμε σε δεύτερη, σε τρίτη, θα έχει καλυφθεί χρονικά το ζήτημα. Τροπολογία 44, άκουσα με μεγάλη προσοχή ε, τις ευαισθησίες, τις αντιδράσεις, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς. Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο συμβαίνει και από πλευράς του συναδέλφου κυρίου Ερτούγκ και πιστεύω ότι η λύση υπάρχει και είναι εφικτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συμβολή σε αυτή τη συζήτηση. Περιμένουμε τις τροπολογίες ε, για να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων προτάσεων. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, τον κάθε ένα και την καθεμία από εσά. Ιδιαίτερα, όπω είπε και ο κύριο Κουμουτσάκο, για τις ε, προτάσεις εκείνε οι οποίες ίσω δεν μπορώ να τι χαρακτηρίσω βεβαίω επικριτικές, αλλά πάντω απαιτούσαν περισσότερα από εμά. Ήταν φιλόδοξε απέναντι στο έργο μα. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά αναφερθώ στα έργα και, και τη μεθοδολογία. Ο κύριος ε, Κουμουτσάκος νομίζω πολύ ξεκάθαρα επεσήμανε ποιος ήταν ο στόχος μας και τι επιδιώκουμε. Εν προκειμένου λοιπόν θα ήθελα και επειδή ακριβώς θεωρώ ότι ορισμένοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εξημών ε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ γιατί βεβαίως Εάν κανεί στη χώρα του, στην πατρίδα του την ιδιαίτερη επικοινωνήσει με τους τοπικούς ε, φορείς ή ακόμα καλύτερα πάει στα Υπουργεία, θα του δώσουν ασφαλώς ένα πακέτο φυλάδια και πληροφορίες, τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητα ορθή ενημέρωση. Γι' αυτό επιδιώξτε περισσότερο καλή ενημέρωση στα κράτη σας, και αυτό το λέω περιλαμβάνοντας και το δικό μου το κράτος, για να δείτε πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, γιατί δεν πρόκειται για τη δουλειά των τελευταίων τριών μήνων, πρόκειται για δουλειά δύο-δυόμιση ετών, που τα κράτη-μέλη ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύτερα κάλεσε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν και στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας αλλά και στην ανάπτυξη των ε, θέσεων και καλό οποιονδήποτε έχει να κάνει επικρίσεις ε, και να ε, απορρίψει κάποιες ιδέες, να ε, τον ελέγξει ως προς τη συμμετοχή του σε αυτή τη φάση της προπαρασκευής. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω επιπλέον ότι εμείς εκφράζουμε το Κοινοβούλιο. Φανταστείτε τι πράττει το Συμβούλιο σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. σε καθοριστική σημασία σημεία το Συμβούλιο, εκεί που πράγματι είναι επώδυνες, επώδυνα τα προβλήματα, εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη για βελτίωση, εκεί που πραγματικά χρειάζεται η αηφορία, το, το Συμβούλιο έχει αποδυναμώσει ουσιαστικά τι θέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τέτοιο βαθμό που θα ήταν καλύτερο να μην υπάρχει καν η πρόταση αυτή. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμεί, ήταν ω Κοινοβούλιο, να αποκαταστήσουμε αυτή την ισορροπία και βέβαια και για λόγου στρατηγικού. Και γι' αυτό σα καλώ να μα υποστηρίξετε. Επίσης, από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφές νομίζω ήδη αν τη διαβάσει κανείς ότι υποστηρίζεται ως μέσο μεταφοράς κατά κύριο λόγο στη διδροτροχιά και η εσωτερική πλωτή οδός. Και εγώ αυτή την προσέγγιση το λέω ρητά, την υποστηρίζω ότι θεωρώ σωστή. Όποιος θεωρεί ότι δεν είναι σωστή, αυτή η λύση βεβαίως ας το πει, δημοκράτες είμαστε, δεχόμαστε τη διαφορετική άποψη, αλλά εγώ προσωπικώς θεωρώ ότι αυτή είναι η ορθή οδός, η ορθή επιλογή. και επίσης για τα CEF και τους δύο συναδέλφους που έχουν αναλάβει τη σχετική εισήγηση. Καλό τους πάντες και τις πάσες να τους υποστηρίξουμε. Είναι μια μεγάλη δουλειά, ένα τεράστιο έργο και πρέπει να τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις έτσι ώστε να κερδίσουν με την υποστήριξη όλου του Κοινοβουλίου την μάχη αυτή. Είπε ο κύριος Κουμουντσάκος ότι τα ΣΥΕΦ είναι ο κινητήρας αυτού του έργου και πρέπει, είναι ο κινητήριος μοχλός και πρέπει να ε, προχωρήσουμε και από αυτή την πλευρά ε, όσο δυνατόν πιο ικανοποιητικά. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύστημα, να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο σύστημα TNT ε, γιατί έτσι πιστεύω πολλοί συνάδελφοι με απορίες σχετικές ιδιαιτέρως ε, με τη χαρτογράφηση, ιδιαίτερως με την γεωγραφική κατανομή κτλ. να βρουν απαντήσεις χάρη στην πρόσβαση αυτή. Γι' αυτό παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να ανοίξει το σύστημα TNT στην πρόσβαση για τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω βέβαια τι θα φέρουν οι λοιπές συζητήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρώτος προθεσμία, σας πενθυμίζω είναι 28 Σεπτεμβρίου και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες 5 ενδεκάτου. Ψηφοφορία 27 αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μικρό διάλειμμα να μαζευτούμε, να ετοιμαστούμε για να υποδεχούμε τους κυρίους Κάλφιν και Μπέγκε για το πολιτισμό δημοσιογραφικό πλαίσιο. Okay, colleagues, if we can go on to the next item on the agenda, which is the exchange of views with our... Με στο επόμενο σημείο, συνάδελφε, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους ηγητές του Κοινοβουλίου ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, με τους κυρίους δηλαδή Μπέγκε και Κάλφιν. Πρώτα-πρώτα, θα πρέπει και τους δύο να σας καλωσορίσουμε στην συνάντησή μας και να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας ε, αναφέρετε ε, τι γίνεται, σε ποια φάση βρίσκονται οι δύο πραγματεύσεις οι οποίες ε, ξεκίνησαν από το άτυπο συνέδριο της Λευκοσίας για τις πτυχές μεταφορών και τουρισμού και όσον αφορά το CF Connecting Euro Facility γιατί θεωρούμε ότι το CEF θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ε, στατικής ανάπτυξης ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε την σημερινή χρηματοοικονομική κρίση. Οπότε, ε, δεν μπορούμε παρά να ακούσουμε με ενδιαφέρον όλα όσα έχετε να μας πείτε, διότι, δεν ξέρω αν είμαι κινδυνολόγος, αλλά πάντως στην Επιτροπή μας φοβόμαστε, φοβόμαστε κάπως ότι το ΣΕΦ με τον Α ή Β τρόπο πρόκειται να περικοπεί ή και να εξαφανιστεί τελείως. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, σας παρακαλώ αν θέλετε να κάνετε τον ακτήριο λάκτισμα όποιος από τους δύο θέλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς τα βρήκατε μεταξύ σας. Ένα δεκάλεπτο καθένας, αν συμφωνείτε. Καλά, ξεκινώ με τον κύριο Κάλφιν. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ ε, στην συνάντηση της ομάδας, διότι θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση που έχουμε μπει, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι συντονισμένο και να έχει μια συνταγμένη θέση όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε τη λέξη διαπραγματεύσεις και αναφέρατε ότι κάπως φοβάστε. Θα μπορούσα να σας ε, απαντήσω ότι εγώ δεν ε, θα συμφωνούσα ακριβώς. Δεν διαλεγόμεθα με το Συμβούλιο, πάντως και εγώ φοβάμαι. Σημίζω με τους φόβους σας γιατί το Συμβούλιο ακόμη πόρο απέχει από το να υιοθετήσει κάποια θέση. Και ξέρετε, πώς αποφασίζει πολλές φορές το Συμβούλιο. Ίσως πρόκειται για κάποιο συμβιβασμό, ο οποίος θα στερείται παντελώς λογικής και συνοχής και συνέπειας. Τέλος πάντων, πριν αποκρισταλώσουμε κάποια θέση, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί οτιδήποτε. Όπως προαναφέρατε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε προσκληθεί εις ε, την συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Ήταν ένα συμβούλιο άτυπο. Έγινε στην Λευκοσία από την ε, Κυπριακή Προεδρία και ήταν μονοθεματικό αυτό το συμβούλιο. Ήταν το θέμα το μονοετές, συγγνώμη το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση. Τα εξής να σας πω τι προέκυψε και να σας πω επίσης και εμείς πώς ε, βλέπουμε τα πράγματα. Τα νέα που προέκυψαν είναι ότι ο πρώτος του Συμβουλίου, κ. Φανρουμπάη πρόκειται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Νοέμβριο. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει στις 22 και 23 του Νοεμβρίου. Οπότε και αυτή η συνάντηση θα συζητήσει μόνο το πολιετές δημοσιομικό πλαίσιο. Γιατί μέχρι τώρα έχει μπει στην ημέρα διαδέξη ποτέ δεν συζητιέται όμω όπω βλέπει και ακόμα και τον Οκτώβριο στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου. Η βασική ιδέα ήταν να συζητηθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα και αυτό επίση ήταν η πρόταση Μπαρόζο όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και το MFF, το πολιετές πλαίσιο, είναι το δεύτερο σημείο Οπότε βλέπετε ότι όταν έχετε πρώτο ένα μεγάλο ευρύτατο θέμα, τότε το επόμενο, το επόμενο εξίσου μεγάλο, αποθείτε και ποτέ δεν συζητείτε όπως πρέπει. Το δε Νοέμβριο πρώτα να έχουμε αυτό το έκτακτο συμβούλιο, το οποίο αποκλειστικά πρόκειται να ασχοληθεί με το πολιτές πλαίσιο. Τι θέλει το Συμβούλιο? Θέλει να προκύψει κάποιος γενικευμένη συμφωνία μέχρι το τέλη του χρόνου, αυτό είναι θετικό γιατί και εμείς θέλουμε να κλειστεί συμφωνία όσο γίνεται συντομότερα γιατί έχουμε μια σειρά νομοθετημάτων και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν και θα πρέπει να ξεκινήσουμε εάν θέλουμε μέχρι τον Ιανουάριο 2014 να έχει εγκριθεί το πλαίσιο. Τώρα, τι άλλα νέα έχουμε χωρίς και με μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ενθουσιασμό, είπε το Συμβούλιο θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ εδώ ως Επιτροπή Μεταφορών. Διότι αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για το ΣΕΦ θα πρέπει να ξεκινήσουν όποτε τυχόν είμαι θα εμείς και το Συμβούλιο έτοιμο. Δεν ξέρω τώρα πώς ε, έχουν ψηφθεί τα πράγματα από τότε στο Συμβούλιο, αρνήθηκαν να συμφωνήσουν μαζί μας για τα θέματα που έχουν σχέση με την απασχόληση, γιατί η κυρία Μπερέ είναι έτοιμη και η Επιτροπή και πρότεινε να αρχίσει ο διάλογος με το Συμβούλιο σχετικός. Το Συμβούλιο όμως αρνήθηκε. Τι δε, περασμένη εβδομάδα έγινε αυτή η άτυπη συνάντηση και συμφωνήσαμε ότι όλα τα ντοσιά πρόκειται να συζητηθούν. Αλλά χωρίς να αποκρισταλωθούν κάποιες αποφάσεις. Έχουμε τώρα δύο βασικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην Κύπρο. Πρώτα πρώτα πώς το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο ε, θα συντονίσουν το έργο τους. Κατά τη γνώμη μου και συμφωνεί και ο συνεισηγητής και το συζητήσαμε είναι ότι οι Υπουργοί δεν θέλουν να διηγούν τα πράγματα σε κάποια φάση ανεξέλεγκτη με όλα αυτά τα έγγραφα, με τι διαπραγματεύσεις ταυτόχρονα και προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στους υπουργούς ότι αυτή η διαδικασία κάθε άλλο παρακτός ελέγχου είναι και οι υπουργοί αν δεν έχουν την εντολή δεν μπορούν να συμφωνήσουν όμως. Και δεύτερον, υιοθετήσαμε την αρχή του ότι τίποτα δεν ισχύει, τίποτα δεν θεωρείται συμπεφωνημένο εάν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα. Αυτά όσον αφορά την έξοδο των διαπραγματεύσεων. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά ανέφεραν ότι οι επικεφαλής των κρατών πρόκειται να επιδρούσουν την προσοχή τους μόνο στα ποσά καταρχήν του πολίτους πλαισίου. Αλλά ίσως και συζητήσουν και τίποτα άλλο. Και πάλι το Κοινοβούλιο είπε ότι και η συνένεση και η συναπόφαση. Έτσι κι αλλιώς το πράσινο φως του Κοινοβουλίου. Και επομένως να ζητηθεί ό,τι θέλουν. Ό,τι τον θέλουν. Αλλά τελικά το Κοινοβούλιο δεν θα συμφωνήσει με τετελεσμένα γεγονότα να θεωρήσει ότι υπήρξε συμφωνία και να μας πούν αυτοί ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμα αυτά. Είπαμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν ήταν επίσημη απόφαση, αλλά τέλο πάντων ακολουθήσαμε αυτή, αυτή είναι η γενική αρχή που είχαμε να ακολουθήσουμε από το Κοινοβούλιο και είπαμε ότι το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να λάβει υπόψη κάποια συμφωνία των επικεφαλής των κυβερνήσεων εάν δεν υπάρξει συμφωνία επί του συνόλου. Και εάν μπορούμε να συνεχίσουμε με τόσο φασιστική θέση. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο συζητήθηκε. Η Κυπριακή Προεδρία παρουσίασε ένα έγγραφο το οποίο αφορά τις διμερείς διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη. Πρέπει να τέψουμε τον χώρο το καλοκαίρι. Είμαι αν δεν έχετε δει αυτό το έγγραφο, εμείς θα σας το δώσουμε. Και πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο είναι μία πρόκληση. Έχουμε εδώ ένα σωρό αποκλειστικές ιδέες, δεν γίνονται όλα αυτά που γράφει και έχουμε επίση και μία σειρά άλλων θεμάτων που τα κατημέλη τα θεωρούν αδιαπραγμάτευτα γιατί λένε για το θέμα που μας καίει ότι από ό,τι φαίνεται αφού δεν υπάρχει συμφωνία για αύξηση του προπολογισμού από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία να συρρυκνωθούν τόσο προτείνει η Κομισιόν. Εγώ δεν έχω δει τέτοιου είδου συμφωνία. Ξέρω ότι είναι διχασμένο το Συμβούλιο. Άρα κάπως υπερβάλλουν. Επίσης λέει εδώ πέρα ότι αν υπάρξουν περικοπές θα υπάρξουν περικοπές για όλες τις πολιτικές. Το κούρεμα που λέμε σε επίπεδο χρηματοκομική σταθερότητα, δηλαδή οριζόντια περικοπή. Δεν θεωρώ ότι βέβαια το κοινοβούλιο, αυτό θα το δεχθεί εύκολα μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο έχουμε πρεσβεύσει είναι ότι δεν δεχόμαστε περικοπές. Και αν τελικά θέλετε να συρρυκνώσετε το προπολογισμό, ε, τότε να κάτσει το Συμβούλιο και να αναθεωρήσει όλες τις πολιτικές και να αποφασίσει με την συρρυγνωμένη πρικοδότηση ποιες προκοπές θα καταργήσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Επίσης, ε, ε, όσον αφορά το ΣΕΦ, ε, υπήρξε μηνύα στο επίσημο έγγραφο και είπαμε ότι τώρα θα πρέπει να καλύψουμε για τις τηλεπικοινωνίες και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να υπάρξει κούρεμα, να υπάρξει διαγραφή, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει γενική συμφωνία δεν είναι οι τηλεπιονίε σημαντικές. Θέλουμε έναν ε, προϋπολογισμό που να μην είναι χαρτί από κάποιο λογιστή, αλλά να, είναι, να έχει όραμα για απασχόληση και ανάπτυξη. Επίσης, είπαν ότι είναι δύσκολοι λοιπόν τα 10 δις από την ε, πολιτική συνοχή να πάνε στο ΣΕΦ. Και αυτό το έγγραφο επομένω θεωρώ ότι αποτελεί μία πρόκληση. Τι επιστροφές είπαν ότι θα καταργηθούν, τα rebates και επίσης να το κοιτάξετε, είναι τρει-τέσσερι σελίδε πολύ ενδιαφέρον αυτό το έγγραφο. Οπότε από πλευρά περιεχομένου είναι διχασμένο το Συμβουλίο. Ο τρόπος να το δείτε, να ότι πρόκειται η Προεδρία να φτιάξει έναν Negotiating Box το Σεπτέμβριο, είπαμε, ίσως θα είναι κάπως καθυστερημένο. Δεν ξέρουμε τι θα πούνε. Υποθέτω δεν θα κάνουν ό,τι και οι Δανείοι όλα να τα βάλουν στο negotiating box. Γιατί αυτό συγχνώνει πάρα πολύ τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να κάνει σωστές διαπραγματεύσεις. Κάτι άλλο τώρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας αναφέρω ότι να πάει. θα, συνεχίσει να προεδρεύει και όπως έχει σήμερα η κατάσταση δεν προβλέπεται κάποιος μηχανισμός για ε, το ποιος θα διαπραγματεύεται από πλευράς του Συμβουλίου. Γενικά ο ομόλογος μας είναι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Άρα αυτό θα ξανασυζητηθεί όπως έχει συζητηθεί επανειλημμένα θα πρέπει πάντως να δούμε ποια είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Το Κοινοβούλιο πάντως πρόκειται να ξεκαθαρίσει ότι η οδήποτε, πρόταση δεν έχει περάσει από τα βούλες μαζί μας δεν την δεχόμαστε. Άρα αυτές είναι οι πιο φρέσκες εξελίξεις από την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βόλφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριος Μπέγκε. Λίγες μόνο παρατηρήσεις. Η ομάδα, η διαπραγματευτική, είναι πολύ ενωμένη και κάθε κρίσιμη για τις περαιτέρω ε, διαπραγματεύσεις πτυχές ε, είναι μέσα στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το πλαίσιο και την πολιτική διαχείριση. Θα ήθελα ξεκινώντας κύριε Πρόεδρε να πω ότι ιδιαίτερα χαιρόμαστε να βλέπουμε τις ομάδες επιφύσης μας, την υποστήριξη, τα σαφή μηνύματα επίσης τα οποία λαμβάνουμε κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Μεταφορών είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία σε σχέση με το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων. Έχουμε πιλωτικά προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσει με την Ουγγρική αρχικά, μετά την Πολωνική και τη Δανική Προεδρία, τώρα υπό Κυπριακή Προεδρία και παλά, παρά το, τα ερωτηματικά για το τι μορφή θα πάρει το τελικό σχέδιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά τα πιλωτικά αυτά προγράμματα. Είναι η πρώτη φορά που αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλήθη να συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων και στην ε, συζήτηση στο πρώτο αυτό στάδιο. Άρα λοιπόν βάλαμε ένα ποδαράκι στην πόρτα και είναι δύσκολο να αφήσουμε πια να κλείσει αυτή η πόρτα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη για να αντιλαμβανόμαστε και πώ θα λειτουργήσει η διαδικασία τη συνένεση για το πολιτέ νομικό πλαίσιο που δεν είναι συναπόφαση. Τη διαδικασία συμφώνη γνώμη, όπου ε, έχουμε επιλογή μόνο να πούμε ναι ή όχι και όχι να αλλάξουμε κάτι. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία που είναι μια, διαδικασία μάθησης θα έλεγα έχει πολύ μεγάλη σημασία και για εμάς και για το Συμβούλιο για να αντιληφθούμε καλύτερα και να προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε καλύτερες διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς αυτούς ε, που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Επίσης είμαστε σε μια κατάσταση και αναφέρθηκε και νωρίτερα, όπου επί δύο ώρες συζητούσαμε θέματα διαδικαστικά. Ε, και ελπίσουμε την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τον κύριο Μαυρογιάννη, τον ε, Κύπριο Υπουργό που θα επισκεφτεί το Στρασβούργο για το πώς θα έχουν τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε μια διάκριση μεταξύ των ε, προγραμμάτων από συναπόφαση και των διαδικασιών και η γραμματεία μας έχει προετοιμάσει το σχετικό υλικό, την τεκμηρίωση για το πού βρισκόμαστε σε επίπεδο συμφωνής νόμης, πού μπορούμε να έχουμε έξω, ε, πέραν του MFF ε, τα σχέδια σε συναπόφαση. Και επίσης από πλευράς μας σαφέστατα λέμε ότι δεν συμμετέχουμε σε προγράμματα, σε έργα συναπόφασης, θα τα πω, απορρίψουμε μόνο για την δική σας αρμοδιότητα, θα τα θα τα απορρίψουμε μόνο, αλλά εάν θεωρείτε εσείς, εσείς όμως ότι είναι χρήσιμο να συζητήσουμε τα ποσά, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, πολύ ευχαρίστω. Προσωπική μου τώρα αίσθηση και χωρίς να θέλω να προκαλέσω ή να επικρίνω το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων. Τώρα που έχουμε διμερείς ε, επαφές, πολύ περισσότερες και ουσιαστικές από ό,τι στο παρελθόν, θα ήθελα να πω ότι βλέπω η ανησυχία του Συμβουλίου των Γενικών Υποθέσεων ως προς την επιτάχυνση των συζητήσεων για τα συναποφασιζόμενα προγράμματα να έχει να κάνει με την ανησυχία τη σχετική με το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο λαμβάνει περισσότερε αρμοδιότητε, παρά τα όσα ορίζει η συνθήκη για τι νομοθετικέ εξουσίε του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και έτσι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό από τι εξουσίε και τι αρμοδιότητε του. Αυτό είναι το ζήτημα που του ανησυχεί και βεβαίω πιστεύω ότι θα πρέπει να διαβάσουν λίγο καλύτερα την συνθήκη τη Λισαβόνα και τα σχετικά, τα σχετικά με τη συναπόφαση σημεία. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι, γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ε, σαφώς δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στις θέσεις της για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τελεία και παύλα, υπήρξαν διαφορετικές θέσεις στο παρελθόν και γι' αυτό υπογραμμίζω τις τοποθετήσεις αυτές, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, για την Κυπριακή Προεδρία και το έγγραφο θέσεων ε, ή ζητημάτων είναι μια μορφή πρόκληση. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δηλώνουν πιο ξεκάθαρα το τι επιδιώκουν και όχι μόνο μείωση 100 δισεκατομμύρια που ζητούν ορισμένα, αλλά και περισσότερες θέσει απασχόληση, ανάπτυξη που διεκδικούν κάποια άλλα, που είναι σημαντικά επίσης ε, και λόγω τη νέα συνθήκη. Και είναι πολύ σημαντικό και εμεί από πλευρά μα να δώσουμε θέσει και με την ενδιάμεση έκθεση από πλευρά του Κοινοβουλίου και να ε, πραγματευτούμε τις θέσεις τους, του Συμβουλίου και τις ανάγκες που εκφράζουν ορισμένα κράτη-μέλη και ενδεχομένως και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές ως προς τα ποσά στον προϋπολογισμό, αλλά και τις πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά και υποχρεώσεις, δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή έχουν αναλευθεί στο παρελθόν από Ευρωπαϊκά Συμβούλια, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, πιστεύω, εξαπαντός να τοποθετηθεί κατά τρόπο σαφή και να μην, ε, για να μην κατηγορηθούμε ότι ε, ξεπερνούμε ορισμένα ποσά, ότι ξεπερνούμε πάντα τα ποσά και ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως πρέπει, αλλά δείχνουμε ότι έχουμε πολιτική υπευθυνότητα και δείχνουμε μια στάση σαφή και στεναρία απέναντι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχαμε λοιπόν ε, καλές παρουσιάσεις, ομιλητές, ένας ομιλητής ε, προσκεκλημένος, ο οποίος εξήγησε πόσο σημαντική είναι η τηλεπικοινωνίες και η ευρύ ζωνικότητα για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν ε, τέλειωσε αυτή η παρουσίαση υπεγράψε στην Κυπριακή Προεδρία ότι θα πρέπει να αλλάξουν στο έγγραφό τους ε, την σχετική παράγραφο για να σημειώσουν τη σημασία της ευρυζωνικότητας. Και σας το λέω αυτό διότι στο Ζαμβούργο, την δεύτερη μου πατρίδα, δεν μπορεί να πουληθεί σπίτι αν δεν έχει και σε μια κάποια περιφέρεια έξω από το κέντρο της πόλης δεν μπορεί να πουληθεί σπίτι αν δεν παρέχει και η υπηρεσία ευρυζωνικότητας, αν δεν είναι εξασφαλισμένο η σύνδεση. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Ε, για τις ενεξελίξεις διαδικασίες θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουμε αρχίσει την επεξεργασία της ενδιάμεσης εκθέσεως. Θα έχουμε ένα πρώτο σχέδιο για τις 14-17 του μηνός θα είναι έτοιμο πιστεύουμε. Πρώτη συζήτηση 19 στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών και για μέλη της Επιτροπής 26 ε, Σεπτεμβρίου και για σας τροπολογίες βεβαίως που εφόσον εξετάσουμε θα ανέξουν ένα επόμενο στάδιο Ενδεχομένω, διόρθωση ή προσαρμογή του προσχεδίου μα, γιατί δεν ξέρουμε στι 24 του μηνό τι θα προκύψει, εάν ενδεχομένω προκύψει νέο έγγραφο για το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων. Θα κάνουν μια προσπάθεια το Συμβούλιο αυτό να προχωρήσει λίγο περισσότερο ε, ή θα αντιμετωπίσουμε καθυστερήσεις ενδεχομένως περισσότερες. Εν πάση μια ευελιξία, μόνο ευελιξία μπορούμε να δείξουμε, ένα αναμονή των εξελίξεων. Όπως είπα, 10-11 Οκτωβρίου αναμένεται η θα αντιμετωπισουμε καθυστερήσει ενδεχομένω περισσότερε. εν στην Επιτροπή των εξελιξεων οπω ειπα 10 11 οκτωβριου αναμενεται η ψηφοφορια στην επιτροπη των προπολογισμων και στην δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου να γίνει ψηφοφορία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εν τέλει με, αυτές τη, με αυτή τη μήνυ ολομέλεια, με την μήνυ ολομέλεια μάλλον. Υπήρχε μια επιλογή. Επίση, υπάρχει μια άλλη προοπτική για ψηφοφορία την τρίτη ημέρα τρίτη τη συνόδου του, του Νοεμβρίου. Αλλά μήπως αυτό σημαίνει σημαντική καθυστόρηση σε σχέση με το Συμβούλιο, μήπω σημαίνει ότι κλείνουμε την πόρτα των διαπραγματεύσεων με την Κυπριακή Προεδρία, γιατί είναι πολύ αργά πια. Ε, μήπω ε, χρειάζεται περισσότερο χρόνος για να ανταποκριθεί στις θέσεις του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, χρειάζεται περισσότερο χρόνος. και οπωσδήποτε ευελιξία. Εν πάση περιπτώσει ευελιξία, αλλά πάντως το σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε ήδη να βάλουμε το πόδι στην πόρτα και να ε, ρίξουμε μια ματιά κλεφτή στα όσα συμβαίνουν από την άλλη πλευρά των διαπραγματεύσεων, των τραπεζών των διαπραγματεύσεων. Αυτά. Και την Πέμπτη στο Στρασβούργο θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να συναντηθούμε για να ενημερωθούμε αμοιβαίω για τι εξελίξει στη διαδικασία του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Προ το παρόν, μπορώ να διαπιστώσω ότι έχουμε ένα καλό σημείο κίνησης, είναι ενωμένο το Κοινοβούλιο, ενιαίες οι θέσεις του και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε πέραν των κάποιων σημείων προς μεταξύ μας στις Επιτροπές να παραμείνουμε ενωμένοι και να επιλήξουμε συν χρόνο το θέμα γιατί μόνο έτσι με ενωμένη στάση δηλαδή μπορεί το Κοινοβούλιο να επιτύχει. 18 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε για όλα αυτά και στην Επιτροπή των Προπολογισμών. Την επομένη θα το έχετε. Δεν θα αργήσει φαντάζομαι. Έχω τώρα εδώ πέρα τους ε, ερωτές. Ρίκε, Αγιάλα, Κάντσα. Ο κ. Σάλλος θέλει το λόγο. Κρατήστε τα χέρια σας ψηλά και θα σας καταγράψουμε. Euh, <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, τοποθέτηση. Διότι εδώ και πάνω από δυο χρόνια δίνει μία σκληρή μάχη μπροστά στις ε, πόρτες των ε, τεθωρακισμένων χρηματοκιβωτίων των κρατών μελών. Σε αυτή την επιτροπή έχουμε σίγουρα ένα σημείο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το Collecting of Facilities αποτελεί και τη μεγάλη μας ευκαιρία δηλαδή να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη και στην καταπολέμηση της ανεργίας και έχουμε έτσι και την ευκαιρία να προχωρήσουμε ε, ε, το σύστημα των υποδομών στην Ευρώπη. Όταν ακούμε τις δυσκολίες, μείωση των 100 δις, το συνολικό φάκελο κλπ. κλπ. Όταν ακούμε δηλαδή όλα αυτά τα καθημερινή, της καθημερινότητάς σας, με αυτά δηλαδή τα 50 εκατομμύρια που βγάλε από το 100 το Συμβούλιο, και ακούμε εδώ όλους να μιλάνε για ανάπτυξη, για καταπολέμηση ανεργίας, για απασχόληση, για πρόοδο. Και όταν έρχονται πια στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και ακούμε τι μας λένε, έχουμε την εντύπωση ότι είναι άλλοι άνθρωποι, άλλες κυβερνήσεις. Εσείς είπατε ότι βασίζεστε στο να ξεκινήσουν οι θεματικές επιτροπές τη συζήτηση με το Συμβούλιο, αλλά πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση ανοίγει χωρίς αριθμούς, χωρίς στοιχεία. Σίγουρα οι θεματικές επιτροπές εργάζονται επί του νομοθετικού ε, φόντου, του νομοθετικού ιστού, αλλά δεν έχουν νούμερα στα χέρια τους. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, με την, ένα μικρό πρόβλημα με την ε, ΡΕΓΙ, την Επιτροπή Περιφερειών. η οποία επίσης ε, γνωμοδοτεί, αλλά έχουμε εντελώ διαφορετική άποψη η μεν με τους δε. Και δεν θέλω να ξεκινήσω εγώ τώρα σίγουρα είναι σημαντικά αυτά τα θέματα, 2,5% κλπ. κλπ. Αλλά έχω την αίσθηση να συμμετέχω μέσα σε έναν εκδιασμό που μου λένε ότι ε, δίνουμε, πλη, δίνουμε παραπάνω. Αλλά μία συγκεντρωτική διαχείριση αυτών των δισεκατομμυρίων θα απέκλειε τις χώρες της συνοχής, γιατί το ποσοστό συγχρηματοδότησης εκτός συνοχής ε, είναι, ε, είναι, είναι σχετικά μικρό. Πρόκειται για δωρεές που είναι πιο ψηλές και από το 50%. Αν αποσύρουμε τώρα εμείς Αν αποσύρουμε εμείς αυτά τα ποσά, τότε θα καταλήξουμε σε μικρά τοπικά έργα. Δεν θα έχουμε αυτά τα μεγάλα δίκτυα. Θα, δημιουργ... θα αφήσουμε απ' έξω τις χώρες της συνοχής δεν θα υπάρξει δυνατότητα. Δηλαδή οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη διασύνδεσης θα αποκλειστούν. Η θέση της ε, Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων παίρνει μια θέση που είναι συζητήσιμη αλλά ξεκίνησαν ένα άτυπο τρίλογο και θα έρθουν στον τρίλογο με μια θέση που σίγουρα θα είναι η θέση του Κοινοβουλίου αλλά η θέση αυτή θα είναι αντίθετη με τη θέση των Επιτροπών Μεταφερών. Τώρα εσείς ε, ως επίτροποι, γιατί και ο κύριος Χάν και ο κύριος Λεβαντόφσκι επενέβησαν προς την ίδια κατεύθυνση με σας, αλλά θα πρέπει εσείς ως επίτροποι να καλμάρετε τα πράγματα. Και θα είναι κρίμα να πάει το Κοινοβούλιο με δύο διαφορετικές θέσεις σε διαφορετικούς ε, ε άτυπους ε, τριλόγους. Ε, θα είναι κάτι το ανεξήγητο. Πρέπει να καταφέρουμε να ξανασυζητήσουμε διότι έχουμε ξεκινήσει παράλληλα, δηλαδή δύο γραμμές που δεν συναντιόνται ποτέ. Το αναφέρω αυτό το θέμα διότι είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, είναι ένα μεγάλο ε, θέμα για την ανάπτυξη και το θέμα των πιστώσεων. Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα συνεχίσω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρικέ. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. κυρίως ε, για αυτά τα μηνύματα πρόοδου που μας δώσατε παρά τις δυσκολίες όπως είπε ο κύριος ε, Μπόγκε. Δηλαδή πρέπει όμως ε, να πείσουμε το Συμβούλιο ότι δεν μπορούμε να λέμε μόνο ναι ή όχι αλλά να έχουμε διάλογο και ανταλλαγή. Το δικό μας πρόβλημα στις επιτροπές δεν είναι μόνο το πρόβλημα με την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων, αλλά είναι το να πάμε σε τρίλογο και να ξεκινήσουμε δηλαδή μία συζήτηση όταν άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές ακολουθούν άλλο δρόμο όταν έχουμε εμείς όλες αυτές τις ανακρίβειες και αμφιβολίες στη γενική θέση. Θα πρέπει λοιπόν να τους καλέσουμε σε τάξη Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε διάλογο όταν άλλοι πηγαίνουν αντίθετα τώρα η Κομισιόν και το Συμβούλιο το ξέρουν ότι άμα αξιοποιήσουμε αυτό το 80% φυσικά και εσείς κύριε Κάλφιν το ξέρετε πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία επίκληση στην τάξη. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω. Για τον κύριο Κάλλας που έλεγε δέκα δις ή αλλιώς εξαφανίζονται. Δεν είπε ότι θα επανερχόντουσαν στο Ταμείο Συνοχής. Εγώ θέλω να ξέρω αν αυτό το ονειρεύτηκα ή είναι πραγματικότητα. Διότι εμείς ε, Εμείς ξέρουμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Ρικέ, ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία, διότι υπάρχει το σκέλος συνοχής ε, που αφορά στη συγχρηματοδότηση για τα δίκτυα. Η Κομισιόν δηλαδή είχε βάλει όλα τα μέσα στη διάθεση όλων ε, για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα σχέδια, ε, τα σχέδια των χωρών συνοχής, να τα διασφαλίσει αυτά τα σχέδια. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή είναι μία ε, θολή απειλή ή είναι κάτι το συγκεκριμένο, δηλαδή αν αυτά τα Αν αυτά τα δέκα δις θα μπουν στο ταμείο, αν αυτά τα 10 δις στο, στο ταμείο ή όχι. Και για το θέμα των συνόρων υπάρχει το πρόβλημα των περασμάτων στα σύνορα που πρέπει να διασφαλιστούν, είναι τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν. Και πέστε μας τι θα, πρέπει, τι θα μπορούσατε να κάνετε. Θα υπάρξει Connecting Europe με αυτή τη χρηματοδότηση που είναι το ελάχιστο κάτω από 10% που χρειάζεται η Ευρώπη για να μπορεί να έχει ένα δίκτυο της προκοπής. Ή αλλιώς ε, το κοινοβούλιο κάνει λάθος. Αυτός είναι ο στόχος. Πώς, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάσνικ. Παρακαλώ, εάν επιτρέπετε ο κύριος Κάντσον θα πρέπει να φύγει. Ε, θέλετε να του δώσετε τη σειρά σας στον τον των ομιλητών. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα λέγατε ναι. Λυπούμε, αλλά εγώ ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να απαντήσω στην προβοκάτσια, στην πρόκληση του Συμβουλίου με κάτι το αντίστοιχο. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι όταν ένα σπίτι καίγεται ή όταν έχουμε μία τραυματική κατάσταση πρέπει να είμαστε σαφείς για το ποια θα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Το ε, θέμα πριν από μια ώρα ήταν η συζήτηση σε αυτήν την Επιτροπή για τα νέα, για τα ε, ΔΕΔ Παύλα μη. Μιλάμε για πολύ μακρόπνοα σχέδια. Στην ε, άλλη η επιτροπή στην οποία συμμετέχω μιλάμε για τα TNA. Ε, όλα αυτά για Όλη αυτή η συζήτηση για τις υποδομές είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα κονδύλια τα οποία διατίθενται, διότι στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει ευρώ. Μιλάω βέβαια σε ορισμένες, για ορισμένες περιοχές μόνο της Ένωσης, αλλά επειδή όμως μιλάμε για έναν κόσμο αλληλεγγύης, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε πιο ευρέως. Λοιπόν, δύο δρόμους έχουμε. Ή εμείς θα πάρουμε αυτά τα λίγα λεφτά και να τα χαρίσουμε τζάμπα, να βρούμε δύο εναλλακτικούς δρόμους για αυτά τα χρήματα, σε μεγάλο βαθμό δηλαδή. Να ορίστε ένα ειδικό μικρό παράδειγμα που δίνει την αρχή του αυτού που εγκρίναμε πέρυσι για το Ταμείο ΕΕΦ για την για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Εμείς εκεί φτιάξαμε ένα μικρό κουμπαρά, ρίξαμε 220 εκατομμύρια και αναπτύσσονται πρώτο, αξιόλογες πρωτοβουλίες και σχέδια, διότι φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να ε, επανέλθουν να γίνουν μάλλον συγκεκριμένες, ας πούμε έχουμε εδώ τις startup οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν, δεν πρέπει να μείνουν στα χαρτιά. Τώρα εδώ έχουμε τρεις κατηγορίες υποδομέγμων. Και θα πρέπει να παλέψουμε ή για να έχουμε τα απαραίτητα ποσά ούτως ώστε να υπάρξουν εκεί επενδύσεις ή αλλιώς να, τα project bonds ως εγγύηση που βγάλαμε εμεί 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό και τα βάλαμε ως εγγύηση για φέτος και του χρόνου, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κάτι το οριστικό μετά το 2014 μέχρι το 2020. Πρέπει να έχουμε εμεί χρηματοδότηση για να δώσουμε αυτές τις εγγύησεις και αυτοί, αυτές είναι οι υποθέσεις Α και F, η υπόθεση Project Bonds και μετά έχουμε και τη θεμελιώδη πολιτική επιλογή να πάμε στην χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη, όχι για να πληρώσουμε τα χρέη ή τις οπισθοχωρήσεις τις αμέλειες, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όταν μιλάμε για τα bond, για τα ομόλογα, να φτιάξουμε ένα πακέτο για την μελλοντική εξέλιξη. Γιατί εμείς εδώ δεν θέλουμε να ομολογοποιήσουμε τα δάνεια πάμε τέλος πάντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ας κάνουμε επιτέλους αυτό το βήμα προς τα μπρον που όλη η Ευρώπη περιμένει δηλαδή για να αρχίσει να προχωράει η οικονομία. Αυτές οι υποδομές είναι απαραίτητες για να μην πεθάνουμε από την ακινησία. Και μετά για να βγούμε και από τη μαύρη τρύπα μέσα από την οικονομική κρίση και να δώσουμε τη λύση. Αυτές είναι οι απαντήσεις στην πρόκληση του Συμβουλίου. Αυτή είναι η αλλαγή πορείας ε, και η αλλαγή οπτικής και λυπούμε αν δεν μπορώ να μείνω. Όπως καταλάβατε, ο Αντών είναι φανατικός οπαδός των ομολογών έργων. Εδώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν τέλειωσε, δεν είχε τελειώσει. Α, θέλεις να μιλήσεις ακόμα. Όχι, έλεγα αν να συνεχίσει, ας περιμένω να τελειώσει. Καλώς λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπέγκε, τον κύριο Κάλφιν που ήρθατε. Πολύ καλό το ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την ε, επισκόπηση και την ε, ενημέρωση πλευρά σα. Είστε οι δύο εισηγητές ε, για τα θέματα αυτά που αφορούν βεβαίως και τις κατευθύνες γραμμές και για τα CEF. Και ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι και εμείς έχουμε δύο συνεισηγητές ε, για, την, για το καθένα από τα θέματα αυτά. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουμε τις δύο αυτές εκθέσεις. Και μεγάλη ενότητα ασφαλώς θα διαπιστώσατε και εσείς και για το TNT και για τα CEF μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Θέλουμε όλοι η εσωτερική αγορά να είναι ένας χώρος που θα περικλεί τον πολίτη, στον οποίο θα δέχει τη θέση του ο πολίτης και θα βρίσκει και το δρόμο για το μέλλον του. Φυσικά μεγάλη σημασία έχουν εδώ οι κοινωνίες, αλλά και οι μεταφορές οι οποίες εκπροσωπούμε εμείς και οι οποίες πιστεύω για πρώτη φορά προχωρούν κατά τέτοιο τρόπο οργανωμένο και ουσιαστικό. Και αυτά τα 50 εκατομμύρια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με νύχια και με δόντια να τα υπερασπιστούμε. Τα 10 δις τα οποία αφορούν τα, τις χώρες συνοχής Ξέρουμε ότι κάποια κράτη θα θέλουν να τα κρατήσουν ως δικά τους κονδύλια σε ένα επιπλέον ε, κορβανά, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλό να μείνουν στην, σε διαθέσιμα έτσι ώστε εκείνοι οι οποίοι τα χρειάζονται να τα αξιοποιήσουν πιο καλά. Και έτσι ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που πράτετε εσείς όχι μόνο για τις υποδομές των μεταφορών αλλά και για το μέλλον της εσωτερικής αγοράς για δε τα ομόλογα έργου που αναφέρθηκαν και νωρίτερα, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει μέσα από τις ε, πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές να προχωρήσει η υπόθεση αυτή για να αποδείξουμε ότι είχε δίκιο όλοι Ρεν, ότι μπορεί τελικά να σηκωθεί η ομίχλη και να δούμε καθαρό ουρανό και μέλλον στην υπόθεση αυτή. Μια σύντομη παρατήρηση εν τέλει. για την ολοκληρωμένη πολιτική για τις θάλασσες που θα εισαχθεί και αυτές τις προτάσεις χρειάζεται λίγο, λίγη βοήθεια, λίγα ποσά, μικρά ποσά, αλλά ξέρουμε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μια μικρή λοιπόν σειρά στον προπολογισμό, αλλά πολύ σημαντική για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τιγά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, διαπραγματευτική ομάδα. Η πληροφόρηση κυκλοφορεί καλά μεταξύ ημών και αυτό είναι πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα της διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και με μας. Εγώ θα ήθελα να επιμένω, επιμείνω σε πολλά πράγματα. Αυτό που είπε ο κύριος Ρικέ, πράγματι Πρέπει να, πρέπει να να μην είμαστε διασπασμένοι μεταξύ μόνο για τις, facilities, για τις connecting facilities με την Περιφερειακή Επιτροπή. Αλλά και συνολικά πρέπει να βρούμε μια κοινή θέση ως κοινοβούλιο ισχυρή και ενιαία. Φιλόδοξη. Ε, πανεθετικά λέω ότι η συζήτηση στο ημικύκλιο θα έχει και επιπτώσεις στην ψηφοφορία. Δηλαδή δεν πρέπει να, να μπει το θέμα στην μήνυ ολομέλεια γιατί το χρονοδιάγραμμα θα στραφεί εναντίον μας. Επίσης, στην έκθεση Σίμψον που θα εγκρίνουμε για, αυτή την, για αυτό το πολιετές δημο, δημοσιονομικό πλαίσιο, θα, ελπίζω να συμφωνήσουμε να εργαστούμε για τη διαλειτουργικότητα παράλληλα και τις ε, διευκολύνσεις παράλληλα με τις connecting ε, facilities, όλους αυτούς τους τρόπους δηλαδή για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσα από τις μεταφορές. Και προγράμματα για διευρωπαϊκά δίκτυα και για τους άλλους τομείς. Μας ζήτησαν να εργαστούμε χωρίς αριθμούς. Το κάναμε αυτό στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για διάφορα προγράμματα. Μετά πρέπει να βρούμε όμως πώς θα λειτουργήσει. Γιατί ξέρουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία προχωρεί με νούμερα. Οπότε και εμείς τότε θα πρέπει να ξαναδούμε τη δική μας στρατηγική. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζήλερ και εγώ πρώτα να ευχαριστήσω τους κυρίους Μπέκη και Κάλφεν για όλα όσα μας είπαν. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια και πρώτα πρώτα κάτι για ένα ευρύτερο πολιτικό θέμα. Το MFF μας πάει στο 2020, δεν είναι μακριά πια. Έχουμε την νέα συνθήκη και έχουμε την... Μας, μας πάει σε μια ε, στις ΗΠΑ της Ευρώπης, για, κάτσουμε τώρα να δούμε. Θα πρέπει να ρίξουμε ματιά πώς καλύπτεται ο προπολογισμό των ΗΠΑ και τι θα πρέπει να γίνει τότε με το δικό μας. Έχουμε την κοινωνική πολιτική, η άμυνα είναι διαφορετικό, αλλά η κοινωνική πολιτική είναι περίπου το 20% του, του ΑΕΠ. Γι' αυτό σας λέω, να σκεφτούμε το MFF στα πλαίσια του του 2020. Οπότε, πώς, πώς θα πάρουν τα ενία της ε, οικονομικής πολιτικής οι Βρυξέλλες και πάλι θα αποτελεί το 1% του ΑΕΠ τον ομοσπονδιακό προπολογισμό. Κάτι άλλο τώρα το οποίο είναι ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας. Το ΣΕΦ, κατά γνώμη μου, εμπεριέχει ένα κίνδυνο. Μας είπατε ήδη για την πληροφορική και αν βγάλετε από τα 50 τα 10 δις, μένουν 40. Η δε πολιτική της συνοχής θα συρρυκνωθεί ενδεχομένως αλλά έχουμε αυτό το 2,5% του ΑΕΠ, άρα λιγότερο όπως παίρνουν τώρα κάποιες χώρες. Να βγάλουμε από το ΣΕΦ τα 10 δις και θα πάρουμε τα ίδια λοιπόν όπως έχουμε στις πρώτη και σήμερα. Όμως, αν πάρετε παραπάνω, άλλα 10 θα μείνουν 30 δις και μετά στο μισό 15. Άρα, τι απομένει, τι θα γίνει το ΣΕΦ, οι χώρε συνοχή, κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν καθόλου την υπόθεση ΣΕΦ ω διάδρομο, γιατί είναι πάρα πολύ, μικρός, πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στη συγχρηματοδότηση. Οπότε το 2020 θα έχουμε μια Ευρώπη λιγότερο συνδεδεμένη. Θα έχουμε μεγαλύτερε ανισότητε μεταξύ κρατών μελών και ιδίω όσον αφορά από τη μία μεριά την περιφέρεια και από την άλλη κεντρική και δυτική Ευρώπη Άρα θα πρέπει να κάτσουμε ως πολιτικοί να σκεφτούμε προσεκτικά την προοπτική του τι θα ισχύσει για το MFF σε μια 7 ετία, 8 ετία από σήμερα. Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό σίγουρα, ο κύριος Ντεμπάγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. εγώ έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις για τους ε, δύο προσκεκλημένους που φυσικά τους ευχαριστούμε που ήρθαν και από τις προηγούμενες ε, παρεμβάσεις καταλάβατε για μας τι σημαίνει το ΣΕΦ. Βεβαίως, ε, ε, το θέμα αυτό συνδέεται και με το προηγούμενο, δηλαδή το δίκτυο των μεταφορών. Εσείς λοιπόν, ως διαπραγματευτική ομάδα ή το Συμβούλιο, οι διαπραγματευτές του, δεν συμφωνείτε ότι εάν έχουν περικοπές στο ΣΕΦ θα πάμε και σε κάποιες συνέπειες για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το TNT. Αν επομένω έχουμε περικοπή της πρικοδότησης όπως πήγε ο Σκάνσιαν, θα έχουμε συνέπειες αρνητικές, θα έχουμε μόχλευση για κάποια καινοτόμα άλλα μέσα πολιτικής. Άρα, ίδια μόχλευση, αλλά τα χρήματα τα οποία τελικά θα εκταμιευθούν θα είναι πολύ λιγότερα. Και άρα, η πρικοδότηση αυτή πόσα προγράμματα θα μπορέσει να καλύψει με αυτά τα 10 δις του Ταμείου συνοχή. Νομίζω ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να μείνουν αυτά τα λεφτά στο ΣΕΦ σύντομα, ε, συγγνώμη, πρόσφατα, το Ελληνικό Συνέδριο δημοσίευσε μια έκθεση όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. Σαφώς προέκυπτε ότι δεν δαπανώνται τα χρήματα όπως θα έπρεπε. Άρα, ακόμα και αν βγάλουμε αυτά τα 10 εκατομμύρια από το Ταμείο και τα φέρουμε στο ΣΕΦ, αυτό είναι λογικό. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα βρούμε και μεταξύ μας εδώ στο Κοινοβούλιο, με την Ρέτζη για παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βγάλουμε χρήματα από την πρικοδότηση του ΣΕΦ, ε, γιατί είναι πάρα πολλές χώρες οι οποίες ωφελούνται και άλλες που θα βρεθούν πιο έμεσα σε όλη την Ευρώπη. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Βέβαια, για μας σε αυτό το ΣΕΦ έχουμε την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία για το γεγονός του ότι ε, όπως είπα δηλαδή δεν ε, εμπιστευόμαστε τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να πούν τι θέλουν αλλιώς δεν θα έχουμε ε, προγράμματα προς τιμές αξίες αλλά θα έχουμε εθνικά προγράμματα να ποιος είναι ο φόβος που είναι σπάθη, η δαμόκλειος που θεωρούμε ότι επικρέματα των κεφαλών μας. Ποιο θέλει τώρα να απαντήσει πρώτος, ο κύριος Μπέγκε ή ο κύριος Κάλφιν. Άντε τώρα, εσείς κύριε Μπέγκε. Ναι, ναι, έχει σημασία ποιος ξεκινάει. Είμαστε τόσο ενωμένοι. Να σας επικοινήσω με τον Δομινίκ Ρικέ. Βεβαίως. Πρόκειται για μια συζήτηση χωρίς νούμερα. Ναι για να αποφύγουμε σε αυτό το χρονικό σημείο να υπάρξει σύγκρουση μέσα στο Κοινοβούλιο και ε, διαφοροποιημένες θέσεις. Από την άλλη, όλοι ξέρουμε γιατί πόσα μιλάμε. Μιλάμε για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των ΣΕΦ, CEF, για τις αρχές της εκθέσεως ΣΟΥΡΟ, 2013 συν 5% ως ελάχιστο δηλαδή για την υλοποίηση όλων των πολιτικών ε, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων και απορρεουσών από τι συνθήκε τη αγώνα. Επίσης, μια φράση που λέει ότι εφόσον το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να διαθέσει τα ποσά αυτά, καλούμε το Συμβούλιο να ορίσει αρνητικές προτεραιότητες για εκείνα τα έργα που θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Γιατί αυτό είναι που δεν αντιλαμβανόμαστε εσύ με το δημόσιο διάλογο, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά και με εξωτερικές σχέσεις, με αναπτυξιακή βοήθεια, με 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και την καινοτομία. Και αν δεν επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, ή μειώσουμε τα ποσά, δεν αντιποκρινόμεθα στις διεθνείς μας υποχρεώσεις για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια 0,7% από το ΕΠ, μόνο δύο τρεις χώρες χρειάζονται για να επιτευχθεί και ως εκ τούτου μας μένει η εξής επιλογή να προσαρμόσουμε τα ποσά έστω να είμαστε αρκετά ειλικρινείς ώστε να δείξουμε να πούμε αυτές και αυτές οι προτεραιότητες δεν θα επιλεγούν και θα καθυστερήσει η υλοποίησή τους. Από την άλλη το Συμβούλιο όλο και παρουσιάζει προτάσεις, ιδέες, δεσμεύσεις, υποχρεώσεις, χωρίς όμως να ενισχύει από την άλλη πλευρά τα ποσά. Δηλαδή αντίστοιχα ενίσχυση των δημοσιονομικών, του δημοσιονομικού σκέλους. Και με την Επιτροπή των Περιφερειακών Θεμάτων έχουμε δει προβλήματα. Mm. Άρα, εάν δεν υπάρξει λύση κατάλληλη στο Κοινοβούλιο, θα πέσουν τα πράγματα, θα περιέλθουν και πάλι στα χέρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πράγμα το οποίο για μένα αποκλείται να είναι καλή λύση ή καλύτερη λύση. Οι επιλογές λοιπόν είναι οι εξή. Είτε συνεννοούνται πρόεδροι, συντονιστές, ε, εισηγητές των επιτροπών, ενδεχομένως και με εμπλοκή της διασκέψης των πρόεδρων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, Ίσως να του βάλουμε όλους μέσα στην ίδια αίθουσα και να κλείσουμε την πόρτα και να τους πούμε θα ανοίξει πόρτα μόνο θα έχετε βρει τη λύση. Η λύση αρχής στην οποία είχαμε καταλήξει ως ε, βάση για την έκθεση Σούρε, ξέρετε ότι ήταν ε, να παγώσουν τα ποσά για την πολιτική συνοχή 2007-2013 και να και το δεύτερο μεγάλο πακέτο Γεωργία στα επίπεδα του 2013. Είναι σαφές ότι ανεξαρτώς της εκβάσεως τα ποσά των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών, υπάρχουν χώρες που ακόμη επιδιώκουν περικοπή της τάξης του 100 εκατομμυρίων. Ξέρετε ότι, υπάρχουν χώρες, ότι δεν πρέπει το Κοινοβούλιο ασφαλώς να οπισθοδρομήσει, να υποχωρήσει σε σχέση με αυτό, μέχρι ότου προκύψει νέα συμφωνία. Αυτό είναι τμήμα και της διαπραγματευτικής μας θέσης και βεβαίως του περιθώριου διαπραγμάτευσης που έχουμε χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να συζητούμε για καινοτόμα δημοσιονομικά μέσα. Ο κ. Κάλντσερ επίση το ανέφερε. Επί παραδείγματα υπάρχει Ταμείο Συνοχής, Ταμείο Εγγύσεων, συγγνώμη, από το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, το οποίο εξασφαλίζει τις ε, δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε τρίτες χώρες κατά δε τις ε, διαπραγματεύσεις των υφισταμένων, των τωρινών δηλαδή πολιτών νοσομικών προοπτικών, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε ιδέες για καινοτόμα μέσα, για την έρευνα και άλλα προγράμματα και είπαμε ότι θα πρέπει όχι μόνο να, όχι να αποφεύγουμε τη συζήτηση και τις διαφωνίες για ένα χαμηλό προϋπολογισμό, αλλά και να επιδιώκουμε να βρίσκουμε νέες ιδέες, γιατί είναι πάνω απ' όλα βέβαια σημαντικό το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε αυτά τα σημαντικά στα καινοτόμα μέσα ε, και να μην χάνουμε και εκτιμένα όπως η συναπόφαση στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Άρα λοιπόν με την απόφαση για τα πραγματικά έργα, με τις εγγυήσεις μπορεί το Κοινοβούλιο να ενταχθεί στον όλο διάλογο για τα μέσα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό είτε είναι κανείς πολύ φιλοευρωπαίος, είτε επιδιώκει μόνο μια εσωτερική αγορά, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ε, τις ε, υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, την ενέργεια που έχουν ουσιώδη σημασία και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη δημιουργία της συνεργασίας. Αυτές λοιπόν οι επιπλέον εναλλακτικέ θα πρέπει να μας απασχολήσουν και βέβαια υπό πολύ συγκεκριμένου όρου και προποθέσει. Κυρία Μάισνερ, νομίζω αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, αν κατάλαβα καλά. Για την πολιτική των θαλασσών, φαντάζομαι θα εννοείται περισσότερο υποδομέ και ούτω καθεξής. Προτάσει υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να συζητήσουμε νομίζω και σαν βάση στους λοιπούς τομείς έρευνας. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μέσο και μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης. Για δε τις επικρίσεις προς την πολιτική συνοχής στη δική μου περιφέρεια. Πολλά έργα μπορώ να σας δείξω που έχουν ε, να παρουσιάσουν ε, κάποια ελλείμματα. Ε, αλλά το θέμα είναι πώς υλοποιούνται τα προγράμματα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο διάθεσης των ποσών. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλά, σωστά αποτελέσματα και ικανοποιητικά ποσά. Είναι επίσης όμως πολύ σημαντικό κατά τη χρονική αυτή στιγμή και όταν έχουμε τη συναπόφαση και το, η συζήτηση για τον προπολογισμό οι διαπραγματευόμενοι να προχωρήσουν σε απλούστευση των κανόνων. Σε αυτό επιμένουμε ιδιαίτερως γιατί ε, δεν μπορώ να δεχθώ το διοικητικό άχθο στου ορισμένου τομεί δραστηριοτήτων, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε πρόκειται για τα κράτη-μέλη, να ενισχύεται σε μία περίοδο προσπάθειας σταθεροποίηση του προπολογισμού το έχω πει και στο παρελθόν, είναι πολύ σημαντικό από τις διαπραγματεύσεις να προκύπτει από γραφειοκρατικοποίηση, μείωση της γραφειοκρατίας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να επιληθέσουμε δηλαδή αν οι κανόνες που έχουμε υλοποιούν ε, τον στόχο της λιγότερης και καλύτερης ε, της λιγότερης γραφειοκρατίας, της καλύτερης διοικητικής ε, λειτουργίας. Και βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε εσωτερικά μεταξύ μας στρατηγικές καλύτερες με βάση και τις δυνατότητες που υπάρχουν για διαπραγματεύσει και πραγματικέ ουσιαστικέ συζητήσει με την Κυπριακή Προεδρία πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μην ε, βρεθούμε εκτό παιδιά. Αλλά προ το παρόν α περιμένουμε την παρουσίαση τη ενδιάμεση έκθεση και τη νομοδότηση. Είδα και τι ε, τροπολογίε πολλών ε, που πολλοί συναδελφοί κατέθεσαν, πολύ σε σχέση με τις πτυχές του πολίτου του δημοσιονομικού πλαισίου Άλλοι μιλούν ιδιαίτερα για τη συναπόφαση. Πάντως η θέση μας θα πάω το ότι είμαστε καταρχήν υπέρ της ενότητας του προϋπολογισμού, καταρχήν, αλλά ταυτόχρονα και καταρχήν τα ποσά αυτά που έχουν βγει τώρα από την πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να ενσωματωθούν ιδάλως προγράμματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το, το Κοινοβούλιο θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα και με την ε, περικοπή των ποσών θα είναι πολύ δύσκολη η υλοποίηση των δεσμεύσεών μας και πρέπει να αποφύγουμε ένα κίνδυνο πάγιο πλέον να υπάρχει μια ε, προηγούμενη δέσμευση η οποία θα λέει ότι θα πάρουμε μόνο 1% περισσότερο επί του ΑΕΠ και βρίσκουμε διμερώς λύσεις για το μένει το δε σχέδιο. Γιατί αν καταλήξουμε σε αυτή τη λύση τότε κινδυνεύει η ενότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, εν γέννη, όχι μόνο για την πρώτη αυτή περίοδο πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά εν γέννη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν 10 χώρε οι οποίε θα υποστηρίζουν ένα σχέδιο και η Επιτροπή θα είναι διατεθειμένη να δεχθεί τι ε, εθνικέ συνεισφορέ, ενώ από την άλλη πλευρά θα προσπαθούμε να αγωνιστούμε για την ενσωμάτωση του Αναπτυξιακού Ταμείου. Πρέπει λοιπόν τα ποσά να επανέλθουν χωρίς να ε, πληγούν οι δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης, CEF και οτιδήποτε άλλο σχετικό. Ευχαριστώ. Κύριο Κάλσιαν. Δεν με τη εμπιστοσύνη σα και των συναδέλφων. Απλώ θα σα πω κάτι το οποίο θίξατε για την προστιθέμενη αξία στη Λευκοσία. Είπαμε και στις δύο πολιτικές ομάδες ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη διάθεση των πόρων της συνοχής. Όμως ε, πω ενδιαφέρον το ότι το ένα εναντίον του Όχι, δεν, οι έννοιε τέλο πάντων πάνε μαζί. Καλύτερη δαπάνηση και περισσότερη συνοχή. Προσθέμενα εξαιρετικά του 27. Και ίσω έτσι θα πρέπει να βλέπουμε και τα του προπολογισμού μα. Διότι για πολλέ χώρε, για όλε ουσιαστικά, του φέρνουν επενδύσει, κρατικέ επενδύσει και όταν μιλούμε για εξυγίανση των εθνικών προϋπολογισμών είναι λογικό το ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα από τα λίγα μέσα που έχουμε για να τονώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία είναι ο προϋπολογισμός ο ευρωπαϊκός. Και είναι πολύ σωστό πράγμα το Making Europe. Σας ευχαριστώ και τους δύο, λέει ο Πρόεδρος, πάρα πολύ για την εισήγησή σας και επίσης για τα όσα ερωτήθηκαν θα κάνουμε και ίσως μια σύντομη συζήτηση στη συνέχεια και όπως είπατε κύριε Μπέγκε η τροπολίες αυτές από ό,τι βλέπω πάνε και εδώ, πάνε και σε, άλλες, και σε άλλα θέματα. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι αυτά που είπατε πρόκειται να αντιγατοπτρίζονται στο κείμενο της δικής μας Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Και ευχαριστούμε και για όλες αυτές τις ώρες που έχετε αναλώσει. Εσείς και οι συνεργάτες σας για τις διαπραγματεύσεις αυτές. με το Συμβούλιο. Με τον εχθρό, όπως τους λέω. Θυμάστε τι έλεγα. Είναι ο κροκόδιλος που ίσα ίσα σκαημίτη από το νερό και όταν δεν το περιμένεις, απέρχεται και σαρπάζει. Ναι, ναι, ναι, μου φαίνεται ότι σωστή παρομοίωση ή μεταφορά τέλος πάντων για το Συμβούλιο. Okay, next item is the Επόμενο τώρα είναι η γνωμοδότηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα ήθελα να εξηγήσω στους αδελφούς ότι λόγω των θερινών διακοπών δεν έχουμε μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες τροπολογίες. Όμως σκέφτηκα, μια που έχουμε εδώ τους δύο συνεισηγητές, να αξιοποιήσουμε την ανταλλαγή απόψεων και να καλύψουμε ό,τι έχουν πει. Τόσο 17 Σεπτεμβρίου, έχουμε την ε, ψυχολογία, έχουμε έτοιμη υπερπλήρη μέση ξέρω Οπότε μα δίνεται σήμερα ευκαιρία μήπω κλείσουμε και κανένα συμβασμό, για την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τέλο πάντων, Πολλέ από τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί από ό,τι νομίζω είναι συμβατέ με την συγγνωμοδότησή μου και κάποιε άλλε νομίζω ότι ασχολούνται με πολύ λεπτομερή θέματα και με κάποια άλλα ζητήματα που όπω είπαμε θα πρέπει να καλυφθούν από την συνήθινη παρασκευαστική διαδικασία και όχι να κολλήσουν στο MFF. Να, να πω ποιε δεν μου αρέσουν. Επίση, θα ήθελα να σα τονίσω το ότι έχουμε την τροπολογία 13 τη δική μου που λέει ότι έχουμε ε, για, για, τις, για ε, τους τίτλους το MFF. Αυτά το χρησιμοποιήσουμε ε, σαν στρατηγική με τους δικούς μας για να μην πέσουμε στην παγίδα του Συμβουλίου. Και βασικά νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε για την νομοπαρασκευαστική διαδικασία, νομοθετική διαδικασία τις λεπτομέρειες για το ΣΕΦ. Θα πρέπει όμως να είναι ευσύνοπτο, ξεκάθαρο το μήνυμά μας για να πείσουμε το Συμβούλιο, αλλά και τους κύριους εμπλεκόμενους εδώ. Και σήμερα προέκυψε από τους δύο εισηγητές ότι χρειάζεται αρκετή πρικοδότηση η οποία με τις σειρά είναι αναγκαία για να τονώσει, να αναθερμάνει την οικονομία, να φτιάξει τις απασχόλησεις, ό,τι θέλετε. Αυτά λοιπόν τώρα έχουμε και κάποιες τροπολογίες τις οποίες δεν συμφωνώ. Ο λόγος είναι ότι δεν, θα, δεν είναι εδώ η θέση τους. Όσον αφορά τώρα την επόμενη εβδομάδα να δούμε αν μπορούμε να κλείσουμε συμβασμό παρά απλώ να διαφωνούμε 2, 4, 7 της κυρίας Αγιάλα έχω πρώτον 5, 11, 23, 24 Ντουράν, Έχω πρόβλημα 9, Ντεμπάκερ 10 και 25, Ντεφεράκεν 20 και 22, κύριο Τασέιρα. Όπως προανέφερα, θα ήθελα πώς και πώς να δω αν μπορώ να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο και μην έχουμε τη σύγκρουση μεταξύ συνήθους νομοθετήματος και MFF. Κατά τα λοιπά, Έχουμε πολλές τροπολογίες. Νομίζω επί των οποίων μπορούμε να τα βρούμε. 14, 31 για το υποτατικό μέσο ή 26 δική μου, Αγιάλας 27, 28 ITS. Μπορούμε κάτι να βρούμε. Επίσης νομίζω ότι κάποιες άλλες είναι χρήσιμες προσθήκες όπως Παρθυμονένα Αγιάλα, 3 Ρίκε, και εξαιτικά ο Ντεμπάκες 17, 19, Μάισνερ, η 30η Φαντάλεν και η Παρθμόν 36, Φιντάντσα, ο Ζιάς και άλλων. Να συμφωνούμε. Συμφωνούμε με αυτές. Ε, ε, αυτή είναι η στρατηγική μου. Και σας επενθυμίζω ότι ψηφίζουμε στις 18 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας. Και όπως ακούσατε στις 18 Οκτωβρίου η Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Θέλει κάποιος κάτι? Εντάξει. Μάλιστα. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτά που άκουσα. Έτσι θα προχωρήσουμε για τις τροπολογίες. Πρόεδρος. Δεν συμφωνώ και από τις τροπολογίες. Γιατί έχουμε τη συναπόφαση που είναι κατά το MFF. Οπότε θα προσπαθήσουμε να τις χτενίσουμε και την επόμενη Στο Στασβούργο ελπίζω να σας κατεβάσω κάποιο πρόταση. Καλά, όλοι εντάξει. Ικανοποιημένοι, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο στο διάφορο. Και σε σας ευχαριστώ όλους και τους ερμηνείς και υπενθυμίζω προσοχή συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.